Dear colleagues. Συνάδελφοι, μου φαίνεται ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Ανακοινώσεις. Σήμερα έχουμε 19 γλώσσες και δεν γίνεται αναμετάδοση. Ναι, we Τώρα, τώρα εν ώψη του διαλόγου με την Κομισιόν καλέσαμε σήμερα τον Επίτροπο Αρία Κανιέτε. Ως συνήθως θα αρχίσουμε με την εισήγηση του Επιτρόπου και μετά τη συζήτηση. Ο κύριος Επίτροπος έχει αμέσως το λόγο. Αμέσως. Honorable members. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω και σας και το Κοινοβούλιο ολόκληρο. Σήμερα θα περιοριστώ στα θέματα που σας αφορούν για φέτος δηλαδή το σύστημα ανταλλαγής εκπομπών energy, the governance of the Union and international climate to towards achieving a climate change agreement in Paris. Με την επικείμενη ίσως αργότερα στο χρόνο συμφωνία στο Παρίσι. Λοιπόν, ποια είναι τα θεμέλια της πολιτικής μας αναχέτησης του διοξιδίου. είναι σημαντικό θέμα για την αναχέτηση των κλιματολογικών αλλαγών. Τον περασμένο Νοέμβριο είχα θελήσει να μεταφέρω σε νομοθεσία τις βασικές αρχές του προγράμματος για την ε, αποδιοξίδωση. Τον περασμένο Οκτώβριο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ζήτησαν σαφείς στόχους από τη βιομηχανία και αλλαγή, ορισμένες αλλαγές. Και μετά το 20 θα συνεχίσουν οι ποσοστώσεις, αλλά λόγω των αδειών που έχουν δοθεί και εξαιρέσεων πρέπει να χρησιμοποιήσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε με περιορισμένο τρόπο και καινοτόμο. για την αναθεώρηση του συστήματος συναλλαγών ε, εκπομπών μετά το 20 πήραμε εκατοντάδες ανταποκρίσεις από πολίτες, λέσχες, επιχειρηματίες κλπ. Ε, μπορώ λοιπόν να σας επαναλάβω σήμερα ότι η αναθεώρηση αυτή θα γίνει μόνο αφού εγκριθεί σχετική νομοθεσία. Ευχαριστώ για την υποστήριξη και του Κοινοβουλίου. Οι διαπραγματεύσεις που γίνονται τώρα πρέπει μάλλον να μπορέσουν μάλλον να καταλήξουν σε ένα σοβαρό συμβιβασμό. Οι διαβουλεύσεις που κάνουμε A lot of work is ongoing to gather all the data from the different sectors, transport, building and mainly agriculture. As you know, the objective is to present legislative proposals in two... Θέλουμε να παρουσιάσουμε και νοπτικές προβουλίες το 2016 και σε ό,τι αφορά τις εργασίες μας για τις οδικές μεταφορές ε, πριν να αναλάβουμε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες ε, θέλω να ακούσω όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη γιατί το θέμα των οδικών μεταφορών και της μείωσης ε, των εκπομπών του άνθρακα είναι πολύ πιο πολύπλοκο από ότι οι υπόλοιποι κανονισμοί. Γι' αυτό θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία για να καλέσω τον Πρόεδρο, τον κύριο Λαβία, για να μιλήσει εκ μέρους της Επιτροπής μας ε, στην διάσκεψη των stakeholders που ε, οργανώνουμε για τις 8 Ιουνίου. Αγαπητοί κύριοι βουλευτές, θέλω να φερθώ σε ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της Ενεργειακής Ένωσης. Θα αναφερθώ στην ενεργειακή αποδοτικότητα που πρέπει να είναι μία από τις κύριες προτεραιότητές μας ε, για να κάνουμε πιο βιώσιμο και φόρο το σύστημα της Ευρώπης. Έχει τεράστιο αντίκτυπο στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα. Θα έχουμε μία ε, στρατηγική για ε, την θέρμανση αλλά και ε, την ψήξη και θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όχι μόνο για να εξοικονομήσουμε χρήματα αλλά και να μειώσουμε τις εκπομπές. Το 2016 θα παρουσιάσουμε και θεώρηση της οδηγίας για την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτό αποτελεί συνέχιση αιτήματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να θεωρήσουμε το 2020 το στόχο έχοντας κατά νου ένα επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 30%. Η αναθεώρηση της οδηγίας ενεργειακής αποδοτικότητας θα ακολουθηθεί από την οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων καθώς αυτό θα ε, μας επιτρέψει να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα. Τέλος, οι πολιτικές ε, ε, για την ενεργειακή αποδοτικότητα σημαίνει ότι η αντικαταστασία στο τομέα της ενέργειας πρέπει να είναι αποτελεσματική πανευρωπαϊκά. Η Κομισιόν ε, έχει αναθεωρήσει αυτές τις οδηγίες τα τελευταία χρόνια. Αυτή η αναθεώρηση δεν βρήκε ότι υπάρχει διείσδυση του οικολογικού σχεδιασμού σε καμία πολιτική. Η πολιτική χέρι υποστήριξη από τα διαφορεμένα μέρη, τη βιομηχανία, ε, τις ΜΚΟ, τους καταναλωτές και έχει πάρα πολλά θετικά Ω ως τις της εξοικονομήσεις ενέργειας έχουμε 465 ευρώ το χρόνο ένα νοικοτηριό και η Θεωρείται ότι δεν χρειάζεται αναθεώρηση για την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού, αλλά θα πρέπει να υπάρχει αναθεώρηση στην οδηγία για την ιδιωτική της θα πρέπει να αλλάξουμε το ΑΑΑ ε, μέχρι το D για να κατανοεί ο καταναλωτής ε, την ετικέτα και να μπορεί να αγοράσει πιο αποτελεσματικά προϊόντα. Επίσης, ε, η εποπτεία της αγοράς και επιβολή θα πρέπει να μειώσουν το κόστος από τη μη συμμόρφωση. Θα πρέπει επίσης να κοινοποιούμε καλύτερα τις πληροφορίες στον πολίτη. Κυρίες και κύριοι, χρειάζεται μεγάλη μεταρρύθμιση των ενεργειακών συστημάτων ε, της Ευρώπης. Αυτό αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να πετύχουμε τους στόχους για την κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση. Η πρώτη προτεραιότητά μου είναι να διασφαλίσω ότι τα κράτη-μέλη σέβονται τους στόχους για τις ενεργές πηγές ενέργειας το 2020 η έκθεση που θα πρέπει να εκδώσουμε φέτος για τις ανανεώσιμες πηγές ε, θα μας οδηγήσει ε, στην επίτευξη των στόχων το 2020. Επίσης προβλέπει η μελέτη ε, ένα πακέτο, μια δέσμη μέτρων για την ανανεώσιμη ενέργεια, για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και βέβαια θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υποστηρίξουμε τις νέες τεχνολογίες και θα έχουμε αλλαγές στην ενεργειακή αγορά εγώ βασίζομαι στην στενή συνεργασία μας γι' αυτό. Το να καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση υπερθυμών ένα σε ανέσουμε πηγές ενέργειας σημαίνει ότι θα υπάρχει και συγκεκριμένη δράση σε άλλους τομείς. Παραδείγματο χάρη, ε, ανακοίνωση για το σχεδιασμό για, για προϊόντα της αγοράς ε, θα είναι κάτι σημαντικό για την καλύτερη ένταξη των ενέσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά θέλουμε να κάνουμε τις αγορές πιο ευέλικτες, διευκολύνοντας μια πιο ενεργή συμμετοχή της αγοράς. Έτσι λοιπόν θα είναι πιο εύκολο έχουμε πηγές να συμμετέχουν στην αγορά επίσης όρις. Αυτό επίσης θα μας οδηγήσει σε μεγαλύτερη έρευνα και τεχνολογία και έχουμε το σχέδιο δράσης για την ενέργεια και τεχνολογία που θα κάνει μία πλήρη ανάλυση των δράσεων που θα αναλάβουμε. Τώρα θέλω να αφαιρθώ στη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης. Όπως ε, ε, υπόθηκε από τους ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων το 2014 και το 2015 η Κομισιόν θα ξεκινήσει μια δυναμική ενέργεια διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης. Θα πρέπει η διαδικασία της κυβερνήσης και παρακολούθησης να διασφαλίσει ότι η δράση σε εθνικό πανευρωπαϊκό επίπεδο συνεισφέρει στους κοινούς στόχους. Αυτή η διακυβέρνηση θα πρέπει να είναι διαφανής που να σέβεται πλήρως τα προνόμια των κρατών μελών. Εγώ δεσμεύομαι πλήρως για να διασφαλίσω ότι θα συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλες τις πτυχές της διακυβέρνησης και φυσικά θέλω να ακούσω τις απόψεις για το πώς να προχωρήσουμε για να ολοκληρώσω. Θέλω να τονίσω τη σημασία του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο να πετύχουμε μια διεθνή συμφωνία φέτο στο Παρίσι για την κλιματική αλλαγή. Η Κομισιόν έχει ε, παρουσιάσει το σχέδιό τη για μια δεσμευτική και φιλόδοξη συμφωνία στο Παρίσι. Θα πρέπει εκεί να περιλαμβάνουμε φιλόδοξου στόχου ε, μείωση των εκπομπών, να διασφαλίζουμε τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Επίση, ε, πρέπει να υπάρχει ε, ενδυνάμωση και αναθεώρηση των των δεσμεύσεων θα πρέπει όλα τα μέρη να παρουσιάσουν σχέδια για τη διευκόλυνση της προσαρμογής και θέλουμε να στείλουμε σαφή μηνύματα στους επενδυτές και να ενεργοποιούμε ε, τη ε, διεθνή δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση. Επίσης ε, πρέπει να έχουμε οικοδόμηση ε, ικανοτήτων για τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, για να αναπτύξουν στρατηγικές χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Ε, τον Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η πρώτη μεγάλη οικονομία που έστειλε την συνεισφορά της στην συνδιάσκεψη των Παρισίων. Μέχρι τώρα μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ρωσία, η Νορβηγία, το Μεξικό, η Καμπών, η Ελβετία και το Λίχτενστάιν έχουν ε, υποβάλει τη συνεισφορά τους για την ε, σύνοδο στο Παρίσι. Μιλάμε για 35 χώρες από τις 198. Ε, έχουμε ένα πολύ μεγάλο πακέτο μέτρων ε, για ε, την κλιματική αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει σε μία οδό προς το να μειώσει κατά 20% τις εγχώριες εκπομπές. Αυτό συνάδει με, αυτό που απαιτείται να μειώσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες τις εκπομπές ε, κατά 85% στο 2050 επίσης ε, αν συγκρίνουμε τα επίπεδα του 2010 σε αυτό πρέπει να φτάσουμε στο 2050 και πρέπει να έχουμε μείωση 40-70% για να πετύχουμε το στόχο των 2 ε, βαθμών Κελσίου εμείς επικεντρωνόμαστε τις προσπαθίες μας ε, στις χώρες που δεν έχουν ακόμη ε, στείλει τα σχέδια αυτά να το κάνουν το συντομότερο. Πολλά πρέπει να κάνουμε τους επόμενους μήνες και η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη-μέλη θα εργαστούν για να διασφαλίσουν ότι είναι στην ατζέντα η κλιματική αλλαγή μέσω δημαρών επαφών και σε πολυμερή φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στείλει αντιπροσωπεία στη διάσκεψη των ε, μερών φέτος. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσει με μία φωνή στη διεθνή σκηνή και οι βουλευτές να συμβάλλουν στο να διασφαλίσουμε για να έχουμε φιλόδοξη και παγκόσμια συμφωνία που θέλει να δει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υψηλή στόχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, από τους 10 πολίτες πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι σοβαρό πρόβλημα και οι 4 από τους 5 πιστεύουν ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να είναι καλή για την οικονομία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και περιμένω να απαντήσω τι ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ Επίτροπε. Τώρα θα αρχίσει ο πρώτος γύρος με τους συντονιστάς. Πίτερ Λίζε πρώτα. Δύο λεπτά ο κάθε ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα με την αφήξή μου. Όπως γνωρίζετε ταυτόχρονα υπάρχει συζήτηση στην Ολομέλεια για ένα θέμα που επεξεργάζεται η δική μας Επίτροπη. Χαίρομαι όμως που είσαστε εδώ Επίτροπε και θέλω να σας συγχαρώ προσωπικά και εξ ονόματος της ομάδας μας πολύ καλά τοποθετηθήκατε ως Επίτροπος για τα ενεργειακά σε αυτά τα θέματα. Ιδιαίτερα βοηθάτε ώστε να υπάρξει μια σωστή τοποθέτηση για ένα πιο φιλόδοξο ε, πρόγραμμα δραστηριοποίησης από πλευράς του Συμβουλίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτον το θέμα διακυβέρνησης, governance. Και εκεί εμπλέκεστε υπέρ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις προσπάθειές σας. Ωστόσο θα ήθελα να ακούσω με κάθε σαφήνεια από εσάς όπου, ότι όπου είναι δυνατόν στην Ενεργειακή Ένωση με οδηγίες και κανονισμούς στη συναπόφαση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου θα προχωρήσουμε και δεν θα υπάρξει καμία οπισθοδρόμηση σε σχέση με για παράδειγμα από ένα κανονισμό να μην καταλήξουμε σε μια διακυβερνητική μέθοδο. Θα ήταν καλό αν το επιβεβαιώνατε αυτό Ρίτα. Δεύτερον, ενεργειακή απόδοση. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιούνκερ πριν από την εκλογή του είπε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ένα ποσοστό 30% θα πρέπει να διασφαλιστεί. Στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση δεν τοποθετείται, δεν υπάρχει τοποθέτηση με τέτοια σαφήνεια. Πώς θα δοθεί η διαβεβαίωση ότι θα γίνει αυτό το υποσχέθηκε ο Ζων Ιούνκερ στο Ευρωκοινοβούλιο. Τρίτη ερώτηση για το εμπόριο ρήπων. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Το carbon leakage, η διαρροή άνθρακα και για την αποθήκευση και όσον αφορά τα, τις θέσεις εργασίας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Συμφωνείτε μαζί μου ότι χρειαζόμαστε σωστές κομμένες και ραμμένες στις ανάγκες μας λύσεις γιατί σε σχέση με το 2008 υπάρχουν επιχειρήσεις που λένε ότι βρίσκονται σε ε, η μειονεκτική θέση. Θα πρέπει να εξετάζουμε σε τακτά διαστήματα αν αυτή είναι η πιο σωστή μέθοδος, σε λεπτομέρειες πάντα. Αληθεύει, πρέπει να δοθεί υποστήριξη, αλλά χρειάζεται μια αναθεώρηση. Ίσως όχι κάθε 10 χρόνια, αλλά σε τακτά διαστήματα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καταρχήν ζητώ συγγνώμη για την απουσία του συντονιστή μας Μάτιας και θα έρθει σε λίγο. Εγώ θα ήθελα να τονίσω το θέμα της θέρμανσης του πλανήτη και η διάσκεψη, τη διάσκεψη των Παρισίων που προβλέπεται για το Δεκέμβριο 15. Σημαντικό και το θέμα της συναλλαγής των αδειών, της εμπορίας δηλαδή των εκπομπών, αλλά όπως και άλλοι συνάδελφοι της ομάδας μας θα μιλήσω και εγώ για αυτό το θέμα πιο εκτεταμένα. Για τη διάσκεψη των Παρισίων και τις δεσμεύσεις της Ένωσης που καταθέσατε στη γραμματεία της, στην 6 την 6η Μαρτίου της διάσκεψης όπως αναείπα και πριν του Παρισίων το Δεκέμβριο. Οι κατευθύνσεις που δώσατε είναι προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί συμφωνούμε ότι πρέπει να επιτραπεί σημαντική μείωση των εκπομπών διοξιδίου κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το 30% σε σύγκριση με το 95% και να αυξηθεί στο 27% στην ενεργειακή μίξη το μερίδιο των ανανεωσίμων για να δώσουμε έτσι το παράδειγμα και σε τρίτες χώρες που φοβούνται να αναλάβουν δεσμεύσεις κατά της θέρμανσης του πλανήτη. Ταυτόχρονα η διάσκεψη αυτή για το κλίμα πρέπει να είναι διάσκεψη όπου θα ληφθούν αποφάσεις, όχι δοκιμαστική. Η διάσκεψη λοιπόν αυτή των Παρισιών παρόλα αυτά δεν είναι αυτός σκοπός αλλά η αρχή, το εναρκτήριο λάκτισμα μιας διαδικασίας που να πείσει την διεθνή κοινότητα να αλλάξει τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή να επιτραπεί αύξηση της θερμοκρασίας κατά λιγότερο από δύο βαθμούς. Αυτό βέβαια θα απαιτήσει και εθνικές δεσμεύσεις κοινούς κανόνες για διαφάνεια και συγκρισιμότητα των δεσμεύσεων και επίσης εργαλεία συνεργασίας που να επιτρέπουν τη μεταφορά τεχνολογίας προς τις χώρες που τη χρειάζονται περισσότερο. Θα επανέλθω τώρα σε ένα θέμα που είναι το πράσινο ταμείο. Ανελήφθησαν δεσμεύσεις στην Κοπεχάγη στη διάσκεψη της Λίμας αποφασίστηκε ένα ύψος 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων αλλά κύριε Πρόεδρε πού βρισκόμαστε τώρα ως προς αυτή τη χρηματοδότηση καθώς και ποια είναι τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα του άτυπου συμβουλίου στη Ρήγα για τους συντηρητικούς τώρα κυρία Διεθνιέσκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να είμαι ευθεία και ειλικρινής. Η Ενεργειακή Ένωση είναι κάτι απογοητευτικό υπό το πολωνικό πρίσμα. Στο παρελθόν ο Ντόναλτ Τούσκ, πρωθυπουργό Πολωνία, είπε ότι η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να βασίζεται σε κοινέ αγορέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο ποσοτήτων φυσικού αερίου. Στο σχέδιο το οποίο κατατίθεται τώρα δεν υπάρχει καμία αναφορά κοινών αγορών και σε σχέση και με τα θέματα του άνθρακα υπάρχουν προβλήματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν τι θα γίνει όσον αφορά τη δική μας ανθρακοβιομηχανία στην Πολωνία στην οποία βασίζεται όλη μας η βιομηχανία στην εκμετάλλευση του άνθρακα. Έχουν πιθανότητα στο μέλλον να επιβιώσουν τα ορυχεία μας μελλοντικά και τι θα γίνει σε σχέση με τις σύγχρονες τεχνολογίες για παράδειγμα για τις υπόγειες δυνατότητες της ε, α, αεροποίησης, ε, του, αεριοποίησης ε, του άνθρακα. Αυτό θα έδινε δυνατότητες, δυνατότητες να διασφαλιστούν θέσεις απασχόλησης σε αυτό τον τομέα και θα μπορούσε να οδηγήσει και σε ωφέλη, σε σημαντικά ωφέλη όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία διότι όλες οι βλαπτικές ουσίες υπό το πρίσμα της καύσης θα αποθηκευόντουσαν υπόγεια. Όμως θα πρέπει να δούμε ότι πόρο απέχουμε από την τεχνολογία αυτή στο να είναι έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί εμπορικά. Θα χρειαζόταν υποστήριξη και συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμποριοποίηση, εμπορευματοποίηση μιας τέτοιας δυνατότητας. Βλέπετε κάποιο ρόλο για αυτή τη τεχνολογία στην Ευρώπη. Δεύτερη ερώτηση. Ανεξέλεγκτες μεταφορές ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ διαφορετικών χωρών που θα μπορούσε να είναι πρόβλημα για την μεταφορά για παράδειγμα από την Βόρεια Γερμανία ή για παράδειγμα μέσω Πολωνίας ή Τσεχίας προς την Νότια Γερμανία πράγμα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στο θέμα των, ε, της φθοράς για παράδειγμα ε, των δικτύων όσον αφορά τα θέματα τεχνολογίας και υποδομών. Τι θα πρέπει να γίνει με τις υποδομές που έχουν ήδη υποστεί βλάβες. Θα μπορούσαν να δοθούν αντισταθμίσεις, ε, να δοθούν κάποιες ενισχύσεις σε όσους έχουν ανάγκη και για την ρύθμιση σε σχέση με την αγορά υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα. Πώς στοχεύετε να ρυθμίσετε αυτό το πρόβλημα μελλοντικά. Θα πρέπει να εμπλακούν σε αυτά τα θέματα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ ο κύριος Κερμπραντή για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επιτροπό Κανιέτε για την πληροφορία πληροφοριών που μας έδωσε σε εισαγωγικές του παρατηρήσεις. Έχω ορισμένες ερωτήσεις. Καταρχήν για το να πετύχουμε τους γενικούς στόχους το 2020. Πάντα ακούμε ότι τα πηγαίνουμε καλά. Αν δω όμως τι συμβαίνει στη δική μου χώρα, είχαμε μείωση για ένα-δύο χρόνια στις εκπομπές μας και τώρα που η οικονομία αρχίζει και πάλι να μεγεθύνεται, είχαμε 1% αύξηση ε, των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Πιστεύετε λοιπόν ότι αυτή θα είναι μια γενική εικόνα για το σύνολο της Ευρώπης Δηλαδή τώρα επιτέλους αρχίζει να μεγενθύνεται η οικονομία εκ νέου. Και δεδομένου αυτού πόσο μακριά βρισκόμαστε με την αποδέσμευση των εκπομπών από την οικονομική ανάπτυξη. Η άλλη ερώτησή μου έχει εμπνευστεί από τις φιλοδοξίες Γερμανίας για το 2040 και φυσικά ξέρουμε όλοι ότι το 2020 δεν είναι το μεγάλο εμπόδιο, είναι το 2050 και το να φτάσουμε εκεί. Μήπω θα ήταν καλή ιδέα να ρωτήσουμε τα κράτη-μέλη, να ζητήσουμε τα κράτη-μέλη να χαράξουν κάποιου χάρτες πορεία για το πώ προβλέψουν να πετύχουν του στόχου του 2050 εν τέλει. Γιατί έχω την εντύπωση ότι εμείς ε, όταν ζοριζόμαστε υποστοχωρούμε και δεν ε, θέλουμε πλέον να λάβουμε τα μέτρα που θα έπρεπε. Έτσι λοιπόν ίσως αυτοί οι οδική χάρτες, σε χάρτες πορείας ε, να ήταν ένα καλύτερο εργαλείο προετοιμασίας και για το Παρίσι. Μια ερώτηση. Είπατε ότι είστε απογοητευμένο για το ότι μόνο 35 χώρες έχουν στείλει τα ένδυση μέχρι τώρα. Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να επιταχύνει τη διαδικασία αυτή. Μπορούμε να κάνουμε κάτι μέσω των χρηματοδοτικών μέσων, παραδείγματο χάρη, και εσεί τι σχεδιάζετε. Ευχαριστώ. Η κυρία Κιλώνα για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Επίτροπο Κανιέτε. Πρώτα, ευτυχώς πρέπει να πω παρατήρησα και είδα ότι η επικοινωνία οι, οι μεταφορές αναφέρθηκαν ως ένα τμήμα και τον Ιούνιο είναι ιδιαίτερα θετικό ότι μια διάσκεψη πρόκειται να διεξαχθεί μια διάσκεψη λέγω πούμε για αυτή τη μικρή σύγχυση που δημιουργήθηκε. Υπήρξε μικροφωνισμός από πλευράς διερμηνίας και υπήρξε πρόβλημα. Λοιπόν, ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό. No, nobody anything. I speak with me. Κανείς δεν αντελήφθη τίποτα σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν. Ε, okay. Ωραία, πολύ καλά. Έστω. Λοιπόν, συνεχίζω. Λοιπόν, συνεχίζω. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Επίτροπο Κανιέτε ότι οι μεταφορές τονίστηκαν ως ένας μη ETS τομέας και στις 18 Ιουνίου <clears throat> θα υπάρξει μια διάσκεψη σχετικά. Ήθελα να ρωτήσω επ' αυτού. Έχει ένα προσωρινό χρονοδιάγραμμα ίσως ο κύριος Κανιέται για αυτό το εγχείρημα. Ποιες απαιτήσει θα τεθούν στον τομέα των μεταφορών σε σχέση με το μέλλον. Και επιπρόσθετα θα ήθελα ταυτόσιμη ερώτηση να διατυπώσω όπως ο κύριος Γκεμπράντη προηγούμενα για τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα, την προστασία του, από τις κλιματικές αλλαγές. Λίγες χώρες, πολύ λίγες χώρες ε, έχουν ε, γνωστοποιήσει τους, ε, τις φιλοδοξίες τους και έχουμε φτάσει ήδη τον, στον Μάιο σχεδόν. Έχουμε φτάσει σε κάποια μέσα που με τα οποία θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενδυναμώσει την πρωτοβουλία αυτή και να τονίσει, να τονώσει την πρωτοβουλία της και τη δράση της. Επίσης και μία ερώτηση θα ήθελα να διατυπώσω για την Ενεργειακή Ένωση. Τι γίνεται ακριβώς, είναι δυνατόν στην Ευρώπη να υπάρξει μια ενιαία τοποθέτηση από πλευρά των Ευρωπαίων με ποιο τρόπο η απεξάρτηση, η ανεξαρτοποίησή μας σε σχέση με τους ενεργειακούς πόρους θα διασφαλιστεί στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πραγματικά για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Και θα θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια ζητήματα, ερωτήματα τα οποία διατυπώθηκαν αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι στις απαντήσεις που θα δώσετε θα υπάρχει και μεγαλύτερη ακρίβεια γιατί ένα από τα μεγαλύτερα μελήματα που έχουμε η ενεργειακή πολιτική και η πολιτική για το κλίμα μία από τις προτεραιότητες δηλαδή της δικής μας επιτροπής επιβάλλεται, επιβάλλεται σε εμά από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου όπου απαιτείται ομοφωνία και βλέπουμε ότι στρατηγικούς προσανατολισμούς δίνει το Συμβούλιο όμως στη συνέχεια το νομοθετικό έργο καλύπτεται από πλευρά συνομοθετικής πρωτοβουλίας Εκεί έχει πρωτοβουλ... δικαίωμα πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η μόνη που έχει τέτοιο δικαίωμα. Και όλο και περισσότερο αποκομίζω την εντύπωση ότι μία από τι προτεραιότητε τη Επιτροπή είναι να ακολουθεί τα όσα λέει και επιβάλλει το Συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, ακούμε ότι θέλει να υπάρξει ο πρόεδρο μια πιο πολιτική επιτροπή. Βλέπουμε όμω στη συνέχεια ότι δεν υπάρχει αυτή η πολιτική επιτροπή και ακολουθεί απλώ τα κελεύσματα του Συμβουλίου. Χρειαζόμαστε μια πιο πολιτική πολιτικού χαρακτήρα, πολιτική επιτροπή και να καταδειχθεί ότι δεν θα ακολουθείτε εσείς ε, πυθύνια τα κελέσματα και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου όταν υπερβαίνουν τα εσκαμένα και όταν πέρα από γενικούς προσανατολισμούς θέλουν να συντάξουν και νομοθετικό έργο στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν. Εσείς, ε, ο Γιούνκερ είχε υποσχεθεί δεσμευτικό στόχο 35, 30% ενεργειακής απόδοσης ε, στις επιδόσεις. Αυτό που αναμένουμε είναι να εκπονηθεί μια νομοθετική πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα τέτοιο δεσμευτικό στόχο 30% και τουλάχιστον προσθέτει ο Κλοντ ελάχιστο, ελάχιστη πρόταση 30% αλλά να έχουμε μια δεσμευτική πρόταση και να μην ακολουθούμε πρωτοβουλίες του Συμβουλίου για τα ανανεώσιμα να είναι η Ευρώπη πρώτη προπομπός και πρωτοπόρος στα ανανεώσιμα δεν είναι όμως δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο αν υπάρχει τέτοιο στόχο στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά όχι στο εθνικό επίπεδο νομοθετικά μπορούμε με πλειοψηφικές πλειοψη... με ψηφοφορίες να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αναμένω μια πιο σοβαρή πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσουμε με τα ανανεώσιμα. Αυτό σημαίνει να δούμε και να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα προχωρούν για τα ανανεώσιμα και όχι μόνο σε ενεργειακό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με γενικόλογους στόχους. Διαφορετικά <clears throat> η πιο πολιτική επιτροπή θα σημαίνει να ακολουθούμε τα κελέσματα του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ο κ. Πετιτσίνη για την τελευταία ομάδα από το FTD. Ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε που ευχαριστούμε που ήρθατε. Εσείς αναφερθήκατε καταρχήν στην έρευνα, ε, στην ε, παραγωγή της ενέργειας. Πέρσι η Κομισιόν δημιουργήσε ένα δίκτυο για την ενέργεια για να συλλέξει και να αναλύσει στοιχεία για τον αντίκτυπο, ε, για το σχιστολιθικό αέριο και για τις τεχνικές εξόριξής του, όπως του φράκινγκ. Και για να δει πόσο δυνατόν είναι να υλοποιηθούν στην επικρατειά μας τέτοια σχέδια εξόρυξης 14 ε, από τα 74 μέλη αυτού του δικτύου είναι υπαλλήλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι υπόλοιπα 60 μέλη, μείον το, 10% είναι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και πάνω το 60% ε, εξυπηρετεί συμφέροντα της βιομηχανίας ε, του φιάκινγκ. Έχουμε 5 διευθυντές από τους οποίους οι δύο εργάζονται στη βιομηχανία συλλογικού ερείου. ένας ε, για ε, την γαλλική βιομηχανία και δύο προέρχονται από κράτη-μέλη που έχουν τεθεί υπέρ, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία. Δηλαδή επιτρέπουμε στην, ε, στον κλάδο, στη βιομηχανία ε, της εξόριξης συστολιστικού αερίου να μονοπολεί τη συζήτηση, ενώ πολλέ φορέ οι πληθυσμοί έχουν τοποθετηθεί κατά. Μπορείτε να μας το σχαλιάσετε. Δεν πιστεύετε ότι η Κομισιόν ε, ε, ε, θα έπρεπε ουσιαστικά να κάνει κάτι απέναντι στη βιομηχανία που προωθεί το φράγκινγκ στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει στην πρώτη δεσμή ερωτήσεων. Thank you, Mr. President. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Λίζε. Σε σχέση με τη διακυβέρνηση την οποία ανέφερε, πρόθεσή μου είναι πλήρως να εμπλακεί και να συμμετέχει το Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλω ένα σύστημα διακυβέρνησης όπου θα παραμένει εκτός το Κοινοβούλιο. Θέλουμε να βρεθεί ένας τρόπος συνεργασίας όπου θα αναλύεται η κατάσταση και θα πρέπει σε σχέση με το Κοινοβούλιο ή τα κράτη-μέλη να υπάρχει δυνατότητα προώθησης γιατί η διακυβέρνηση είναι η μόνη δυνατότητα να μπορούμε να επιτύχουμε την ευθυγράμμιση είτε πρόκειται για τις εκπομπές ρήπων είτε για τα ανανεώσιμα είτε για την ενεργειακή αποδοτικότητα και απόδοση και σε όλες τις παραμέτρους της ενεργειακής πολιτικής η διασύνδεση του συνόλου αυτών των παραμέτρων είναι σημαντική. Προσπάθειά μου πρέπει να είναι το Κοινοβούλιο να συμμετέχει στην δυνατότητα δημιουργίας ενός συστήματος διακυβέρνησης μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου γι' αυτό. Για την ενεργειακή αποδοτικότητα είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε και το είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ ότι θέλουμε 30% με δεσμευτικούς στόχους να προχωρήσουμε σε αυτή την παράμετρο. Απαντώντας προς ε, την παρέμβαση ΕΚΟΤ Φυσικά είναι ανεξάρτητη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει το δικαίωμα ανάληψη πρωτοβουλία και λαμβάνει υπόψη να η Επιτροπή αυτά τα οποία λέγει το Συμβούλιο και όταν υπάρχει ομοφωνία και υπάρχει κάποιο συμπέρασμα πρέπει να επεξεργαζόμαστε την δυνατότητα συνέχισης της πορεία. Μπορούμε και να εισακούσουμε και το Κοινοβούλιο. Πρόθεσή μας είναι όμως ε, να μπορούμε να συνεχίζουμε με την πρόθεση του ε, Προέδρου Γιούγκερ με αυτή τη βάση. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε ξεκινώντας ε, για παράδειγμα το έργο μας, να μπορέσουμε με αυτή τη βάση να προχωρήσουμε. Τώρα για την διαρροή άνθρακα. Για την διαρροή άνθρακα αυτό που κάναμε τι είναι. Είναι συναντηθήκαμε είχαμε μια συνάντηση με τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υποβάλαμε ένα ερωτηματολόγιο μέσω του οποίου προσπαθήσαμε να υπάρξει μέσω μιας κοινή προσέγγισης των απαντήσεων η κοινή εκπόνηση μιας κοινή απάντησης και ρύθμισης από πλευράς μας για τη ρύθμιση διαφόρων τομέων ε, υπό το φως των ε, γεγονότων, ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν με την μεθοδολογία επιμερισμού ώστε να υπάρξει ένας, ένα αποτελεσματικό πλαίσιο. Δεύτερον, οι τιμές που θα πρέπει να αναπροσανατολίζονται σε ποια βάση, κάθε αναέτος κάθε δύο ή τρία χρόνια ή σε πολιετή διαστήματα. Ποια θα είναι η πιο σκόπιμη μέθοδος ε, για να μπορέσει να ε, βελτιωθεί η μέθοδος ε, αυτή με συλλογή στοιχείων και την αξιολόγησή τους με τις βέλτιστες προδιαγραφές. Τι θα πρέπει να γίνει σε σχέση με την παραγωγή αυτών των στοιχείων. 5. Ποιες αλλαγές θα προτείνατε στις διαρροές, στο πρόβλημα διαρροής άνθρακα θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει την προσέγγιση δύο διαφορετικών ε, ομάδων σε σχέση με την διαρροή άνθρακα διότι εδώ υπάρχουν ασύμετροι παράγοντες για παράδειγμα για τη μία ομάδα και σε σχέση με την ε, προσέγγιση αυτή για τον επιμερισμό τομέων για το τομείς υψηλού κινδύνου να υπάρχει επιμερισμός ε, σε δύο ή σε τρεις και περισσότερες ομάδες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων διαρροής άνθρακα και πώς θα πρέπει η διαφορετική εμπλοκή διαφορετικών τομέων να αντιμετωπιστεί. Τους ρωτήσαμε λοιπόν, υποβάλαμε αυτό το πλήρες ερωτηματολόγιο για να προσπαθήσουμε να δούμε αν θα μπορούσε να υιοθετηθεί μια κοινή ε, προσέγγιση. Φυσικά θα υπάρξουν κάποιοι ε, τομείς ε, που κάποιους, από αυτούς, κάποιες από αυτές τις πτυχές θα μπορέσουν να τις εντάξουν και να ευθυγραμμιστούν. Είμαστε πρόθυμοι να λάβουμε και να εξετάσουμε οποιασδήποτε ε, απόψεις και προτάσεις ε, κατατεθούν και θα τις αναλύσουμε και αυτό κάνουμε. Αφού γραζόμαστε τις απόψεις των εμπλεκομένων, των stakeholders, ακούμε τις απόψεις τους, αναλύουμε όλες τις απαντήσεις και μετά θα επανέλθουμε το δυνατόν ταχύτερο με τις προτάσεις μας για τη ρύθμιση του τομέα αυτού. Απαντώντας τώρα στον κύριο Περνόν, είναι σαφές ε, ότι το Παρίσι θα είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα. Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών με 198 κράτη που θα πρέπει ομόφωνα να αποφασίσουν και εδώ δεν έχουμε θέμα ομοφωνίας αλλά ε, ειδικής ε, πλειοψηφίας αυτό περιπλέκει τα πράγματα, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να δραθούμε σε ευκαιρία και να σημειώσουμε επιτυχία. Είναι κάτι σημαντικό αυτό το οποίο επισημάνατε. Το Παρίσι δεν είναι το τέρμα της διαδρομής. Έχουμε καθορίσει τον καθορισμό των στόχων, την διαφάνεια, την λογοδοσία, την εποπτεία, μια δυναμική διαδικασία προώθησης και για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν στη Λίμα, ενώ δεν καταφέραμε στη Λίμα του Περού να πετύχουμε ιδιαίτερα σε σχέση με την Κίνα που δεν ήθελε μια αξιολόγηση αυτού, αυτής της διαδικασίας με την ποσοστοποίηση των επιπτώσεων όλων αυτών των παραμέτρων προτού καταλήξουμε στο Παρίσι γι' αυτό αποφασίσαμε να διοργανώσουμε Οκτώβριος δεν είναι μια διάσκεψη που θα προσκληθούν όλες οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, και οι κοινοβουλευτικοί πρόσωποι να προσέλθουν στο Μαρόκο και να αναλυθούν όλες οι παράμετροι και το επίπεδο φιλοδοξιών των προτάσεων. Ίσως μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια άλλα στοιχεία και όχι στους δύο βαθμούς για παράδειγμα. Ε, και αυτό θα ήταν ένα μήνυμα το οποίο θα αποσταλόταν ότι πρέπει να θεσπιστεί μια περιοδική σε τακτά διαστήματα αναθεώρηση ή μεταρρύθμιση ώστε το 2050 να μπορούμε να έχουμε καταλήξει σε ποσοστοποίηση αποδοτική και αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Αναφερθήκατε στο θέμα ποιες χώρες θα συμφωνήσουν με το Κλιματολογικό Ταμείο, το Ταμείο για τις Κλιματικές Αλλαγές. Κάποιες χώρες δεσμεύουν μεγαλύτερα κονδύλια. Αν δείτε τον ετήσιο προϋπολογισμό, τους ετήσιους προϋπολογισμούς, δεν είναι επαρκή τα κονδύλια, δεν είναι τα κονδύλια διαθέσιμα. Και ακόμα και υπάρχουν κοινοβουλευτικοί που έχουν επιφυλάξεις. Έχουμε ένα συνολικό ποσό 10 δισεκατομμύριων, δισεκατομμυρίων δολαρίων ακόμα και σε σχέση με το Περού μικρή αυτή η εμβέλεια αυτού ποσού και σε σχέση με τις είπα το πρόβλημα ποιο είναι τώρα ότι πρέπει και χρειαζόμαστε να μπορέσει να, να αρχίσει να λειτουργεί σε χρηματοοικονομικά σχέδια και προγράμματα. Αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να επιληθούν όλα τα προβλήματα στο που έχουν τεθεί στο τραπέζι ώστε να υπάρχει μια αυθεντική δυνατότητα για τις αναπτυσσόμενες χώρες να αναγνωρίσουν ότι έχουν ένα αυθεντικό εργαλείο στα χέρια τους, ένα μέσο να προχωρήσουν με αυτό το μέσο που έχουμε δημιουργήσει και από πλευράς ε, των, της, ε, των βιομηχανικών κύκλων και της υποστήριξης που έχει, έχουν δώσει σε αυτή την πρωτοβουλία για έγκριση καταφέραμε τελικά να καταλήξουμε σε αυτό το βαθμό συμφωνίας, όχι όμως χωρίς ε, δυσκολίες. Κάποια κράτη-μέλη ήθελαν να περάσουμε πάνω από το 40% άμεσα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η χρήση των γεών, η αλλαγή χρήσης γεών και το τι θα γινόταν σε σχέση για παράδειγμα με το 40% ή την μείωση του 40% και ε, ετίθετο προβλήματα για κάποιες χώρες και πάλι καταλήξαμε να ε, προχωρήσουμε στο να επιτευχθεί μια συμφωνία και εγώ πιστεύω ότι το πιο φιλόδοξο που έχουμε ενώπιον μας αυτή τη στιγμή είναι αυτό αλλά έχουμε και άλλα θέματα που πιστεύω ότι για παράδειγμα ο κ. Γκεμπράντη το ανέφερε δεν είναι και είπε ότι ότι αληθεύει ότι ένας περιορισμένος αριθμός κρατών της λέσχης των 7 της ομάδας G των 7 ή της λέσχης των 20 ε, προχώρησαν. Θα πρέπει όμως έγκαιρα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ώστε αυτό να αποτελέσει κίνητρο για τις υπόλοιπες χώρες να προχωρήσουν και εκείνες. Εργαζόμαστε με αυτή την ομάδα τη λέσχη των 7 και των 20 για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε σχέση και με συνάντηση του Αμβούργου και με την ομάδα του Πέτερσμπεργκ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να δώσουμε την, ε, το μήνυμα ότι όλα τα αναπτυγμένα κράτη θα πρέπει να προχωρήσουν. Είχα πάει τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον σε ένα τέτοιο φόρουμ, σε ένα τέτοιο βήμα και η Κίνα και η Αυστραλία, μεγάλες χώρες δηλαδή, έστειλαν το μήνυμα ότι είχαν την πρόθεση να προσχωρήσουν και άλλοι θα το κάνουν αυτό λίγο αργότερα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Πρέπει να συνεργαστούμε με τις αναπτυσσόμενες χώρες για να τις βοηθήσουμε να προχωρήσουν. Δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να προετοιμαστούν αυτές οι χώρες και να τις συνδράμουμε. Επίσης το για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις κοινέ αγορές ε, φυσικού αερίου που δεν προχωρήσαμε είπατε το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα πλαίσιο πενταετές για μια τέτοιου είδου στρατηγική. Δεν υλοποιούνται όλα άμεσα κατά το πρώτο έτος λειτουργίας. Υπάρχουν, υπάρχουν ανάγκες να προετοιμάσουμε κάποια παραμέτρους ώστε να μπορέσουν να οριμάσουν και να εξελιχθούν μετά. Τώρα, σε σχέση με την τροφοδοσία μας με φυσικό αέριο, πρέπει να δούμε για παράδειγμα με το σχέδιο ε, άμεσης αντιμετώπισης αναγκών ή κατεπίγουσας αντιμετώπισης αναγκών. Το τι θα γίνει με το φυσικό αέριο. Όταν εξαρτάται μια χώρα από έναν πάροχο μόνο ή σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο υποχρεώσεων ο, ο ρόλος του, των κανόνων του ανταγωνισμού, ο ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αναλυθούν και θα γίνουν όλα αυτά όταν θα έρθει η ώρα να προχωρήσουμε με αυτή τη μεταρρύθμιση. Μετά, το ερώτημα το οποίο τέθη ήταν ε, το πρόβλημα του άνθρακα που τέθηκε από την Πολωνία. Ο άνθρακας θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ενεργειακό μείγμα πηγών ενεργειακών της Ευρώπης. Έχει καθοριστεί σαφώς ότι κάθε χώρα, κάθε κράτος μέλος έχει κυριαρχικό δικαίωμα να αποφασίζει το ενεργειακό της μείγμα. Όμως οι χώρες έχουν επίσης την υποχρέωση να σέβονται τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς εκπομπών αερίων. Και αυτό είναι ένα άλλο σκέλος που πρέπει να είναι σεβαστό. Θα βοηθήσουμε όσο είναι δυνατόν από πλευρά μας ώστε σε σχέση με τα όσα αναφέρονται για τη διαρροή άνθρακα και σε σχέση με την υποστήριξη ε, προγραμμάτων και δυνατοτήτων επιχειρησιακών να βοηθήσουμε ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καύσης ε, που δημιουργούν προβλήματα στις χώρες αυτές και να βοηθηθούν οι χώρες αυτές. Αυτή είναι μια λύση, αυθεντική λύση. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε την Κίνα, τη ΣΥΠΑ, ώστε να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε αυτό το μείγμα και να είναι αποτελεσματική η πολιτική μας με αυτή την τεχνική τεχνολογία και την χρήση των δυνατοτήτων χώρες που δεν είναι δυνατόν να είναι αποτελεσματικές αυτή τη στιγμή με την ε, αντιμετώπιση διοξιδίου του άνθρακα πρέπει να δούμε πώς μπορούν να δημιουργήσουν δίκτυα ασφάλειας και να βοηθηθούν. Αυτό θα απαιτήσει βέβαια θα απαιτήσει συγκεκριμένες ενέργειες δεν θα είναι εύκολο θα πρέπει όμως να συνεχίσουμε τις επενδύσεις μας επενδύοντας σε αυτό το εγχείρημα και να προσπαθήσουμε λαμβάνοντας υπόψη το ότι κάποιες χώρες βρίσκονται είναι πιο προηγμένες από κάποιες άλλες και έχουν λιγότερα προβλήματα με αυτή τη διαφοροποίηση να δραστηριοποιηθούμε. Αναφερθήκατε στις ροές ηλεκτρικής ενέργειας για τα δίκτυα. Μια πολιτική πρέπει να ακολουθηθεί για την διασύνδεση των υποδομών και πρέπει και για τον ηλεκτρισμό αυτό να μπορέσει να γίνει. Δεν έχουμε φτάσει στο 10% του 2020, ούτε ακόμα φυσικά στον πολύ πιο φιλόδοξο στόχο του 2030. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν την προσπάθεια για τη διασύνδεση αυτή. Και τέλος, ρωτήσατε ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, ρύθμιση των αγορών. Πρέπει να σεβόμαστε τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ε, ΡΑΕ ε, ενέργειας. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη και τις ανάγκες που υπάρχουν μεταξύ χωρών ώστε σε περιφερειακό επίπεδο ή σε διαμεθοριακά ε, ζητήματα να υπάρχει ένας Ευρωπα... Ευρωπαίος ρυθμιστής, μια Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή που θα διαμεσολαβεί μεταξύ των ε, εθνικών ρυθμιστικών αρχών και έτσι θα εντάξουμε την αγορά σε ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Κύριο Κεμπράντη ρώτησε, έθεσε μια πολύ δύσκολη, ακραίως δύσκολη ερώτηση. Ποια είναι η γενική εικόνα των στόχων σφαιρικά η εικόνα των στόχων που έχουμε θέσει είναι ότι φαίνεται ότι είναι εφικτή και μπορούν να επιτευχθούν ε, οι στόχοι αυτοί. Όμως ένας δημιουργεί κάποια προβλήματα, η ενεργειακή αποδοτικότητα. Με αυτό το στόχο αυτή τη στιγμή οι προοπτικές τι δείχνουν. Δείχνουν 18,5% θα βρεθούμε κοντά στο στόχο με τις σημερινές πολιτικές μας. Αν γίνει κάτι παραπάνω από τα κράτη-μέλη, ίσως θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο 20%. Αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλίσω ότι όλα τα κράτη-μέλη θα εφαρμόζουν τις διατάξεις για την ενεργειακή αποδοτικότητα στην ε, ε, δράση τους ε, και σε σχέση με πολλά κράτη-μέλη πρέπει οι δικές τους δράσεις να οδηγούν στην εφαρμογή αυτών των διατάξεων και ε, ρυθμίσεων. Έχουμε αναγνωρίσει ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα λόγω της αύξησης των οικονομικών δραστηριοτήτων ε, σημείωσε αυτή την εξέλιξη. Τώρα ανακάμπτουμε με ένα βραδύτερο ρυθμό. Η τελευταία φάση για το 2020 θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Το να πάμε από το 20% στο 30% θα είναι πολύ πιο δύσκολο ή από το 2020 στο 2030 θα είναι δύσκολο εγχείρημα και θα πρέπει εδώ να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε για να επιτευχθεί ο στόχος με, με το πρόγραμμα, το σχέδιο ε, για ένα πρόγραμμα στήριξη σταθεροποίησης της ενεργειακής αποδοτικότητας κάτι που θέλει και το Κοινοβούλιο να επιτευχθεί το διάβασα ναι για τη δυνατότητα των κρατών μιλών να, να θεσπίσουν ένα σύστημα. Καταρχήν θα πρέπει να θέσουμε το νομοθετικό πλαίσιο για να πετύχουμε τους στόχους του 2030 και κατόπιν θα σκεφτούμε τι θα γίνει. Γιατί καταρχήν πρέπει να έχουμε ρυθμιστική ασφάλεια. Τα κράτη-μέλη πρέπει να ξέρουν ε, ε, ότι ισχύει η νομοθεσία σε όλα για το ETS, ε, για την ενεργειακή αποδοτικότητα και όταν θα γνωρίζουν τους κανόνες που θα ισχύουν, τότε θα δούμε πώς μπορούμε να καταρτήσουμε δικό χάρτη. Γιατί ναι, έχουμε ε, ένα στόχο στο Παρίσι για το 2050, αλλά ε, καταρχήν το πρώτο τμήμα της οδού φτάνει μέχρι το 2030. Μέχρι εκεί είχε σχεδιάσει η Κομισιόν, αλλά φυσικά θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για το μέλλον. Δίκιο έχετε λοιπόν. Και τελευταία ερώτηση. της ε, κυρίας Για τις μεταφορές μου θέσατε μια ερώτηση. Αν ε, και ο κύριος Έκοτ ε, θα πει ότι ακολουθώ τη θέση του Συμβουλίου, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Οκτωβρίου μας έλεγαν ε, ότι οι μεταφορές ε, θα μπουν στο τμήμα μη ETS, σύστημα εμπορίας εκπομπών. Εμείς ε, εργαζόμαστε για τη μεταρρύθμιση του μελλοντικού συστήματος εμπορίας εκπομπών και θα συμπεριλάβουμε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις μεταφορές, τη γεωργία και τα κτίρια. Τα συμπεράσματα επίσης υπενθυμίζουν ότι οι μεταφορές μπορεί να συμπεριληφθούν στο ETS της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κανένα κράτος μέλος δεν το έχει πράξει ακόμη. Και η Κομισιόν είναι έτοιμη φυσικά να βοηθήσει συμπεριλαμβάνοντας ε, τις μεταφορές ε, ε στο e της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά θεωρούμε ότι είναι κάτι πολύπλοκο και πρέπει να το συζητήσουμε παραπέρα. Και δεν νομίζω ότι η συμπερίληψη των μεταφορών μπορεί να αντικαταστήσει ε, τα πρότυπα της ε, εμπορίας εκπομπών. Θα είναι κάτι συμπληρωματικό, αλλά δεν θα αντικαταστήσει τα πρότυπα των εκπομπών. Τι περαιτέρω μπορούμε να κάνουμε για να αναχαιτήσουμε την κλιματική αλλαγή. Έχουμε την κατάρτιση ενός χάρτη με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ε, έχουμε επαφές με Κίνα, Αυστραλία, Καναδά και άλλες ε, χώρες στο Οικονομικό Φόρουμ και φυσικά και με την Ινδία που είναι μια πολύ σχετική χώρα αλλά και η Βραζιλία για να τις ε, παραπείσουμε να παρουσιάσουμε τις εθνικά Καθαρισμένες προθέσεις εισφοράς το γρηγορότερο, τα indices και επίσης για την ενεργειακή ένωση, τι θα κάνουμε για τα κτίρια. Εμείς ε, εργαζόμαστε προς την ανεξαρτησία, κυρίως για το αέριο. Έχουμε έξι χώρες που βασίζονται σε ένα και μόνο προμηθευτή. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κάνουμε πολλά. Καταρχήν να αναπτύξουμε το νότιο διάδρομο για να αναπτύξουμε το διάδρομο μέσα στο Αζερβαϊτζάν. Έχουμε διάλογο με πολύ σημαντικές χώρες ε, στο μέλλον όπως η Αγγελία και θέλουμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας και με την Ορβηγία αλλά θα θέλουμε και να έχουμε και μια στρατηγική υγροποιημένου φυσικού αερίου για να έχουμε μια εναλλακτική για τους αγωγούς που χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Κούτ. Το Συμβούλιο θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι η ανάπτυξη του πακέτου 2030 θα πρέπει να γίνει με ομοφωνία. Ξέρετε όπως αυτά τα θέματα υπόκειται σε ειδική πλειοψηφία και η Κομισιόν έχει το δικαίωμα ανάληψης πρωτοβουλία. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε να είμαστε στην δυνατόν πιο και να σεβαστούμε τους συμβιβασμούς ε, του κυρίου Γιάνκερ ε, στις ομιλίες του. Στις ομιλίες που εκφώνησα και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τέλος. Υπήρχε και άλλη μια ερώτηση για το θέμα της ηγεσία στο ότι πρέπει να υπερισχύσουν οι ενώσιμες πηγές ενέργειας. Φυσικά πρέπει να αλλάξουμε την οδηγία και αποκοινούμε τη διακυβέρνηση θα πρέπει ε, να έχουμε μια σαφή διαδικασία για να διαπιστώνουμε το επίπεδο της πρόοδου. Αλλά πρέπει και να δημιουργήσουμε ε, δυνατότητες ε, και ανάπτυξης τεχνολογίας ε, μέσω των κατάλληλων ταμείων και να βάλουμε τη δυνατά μα για να διευκολύνουμε τη συμπερίληψη των ενώσιμων πηγών ενέργεια στο δίκτυο. Γιατί αυτή, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τις ΑΠΕ είναι η έλλειψη διασυνδεσιμότητας ε, μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό είναι σαφές πρόβλημα. Έχουμε πρέπει να κάνουμε όλες τις διασυνδέσεις και πρέπει να εναρμονίσουμε ε, ότι η υποστήριξη για τις ανανεώσιμες προσανατολίζεται περισσότερο στην αγορά και δεν προκαλεί στρεβλώσεις. Και θα πρέπει, και μάλλον πρόκειται να παρουσιάσουμε πριν από το καλοκαίρι, μία ανακοίνωση για το σχεδιασμό της ενεργειακής αγοράς Εκεί θα καθορίσουμε πώς θα διευκολύνουμε τη συμπερίληψη των ανανάσιμων πηγών στο Γενικό Σύστημα Ενέργειας. Κύριε Πεντιτσίνη, αναφερθήκατε στο συστολιστικό αέριο. Τώρα προβαίνουμε στη χαρτογράφηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ξέρουμε πού ακριβώς ε, έχουμε πραγματικές καταστάσεις, πού έχουμε διαθέσιμο σχιστολιθικό αέριο αυτό και αφετέρου η τεχνική πλατφόρμα που προσπαθεί αυτή τη στιγμή να αναλύσει τις διάφορες καταστάσεις να δίνει συμβουλές στην Κομισιόν. Η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει μια απόφαση όταν θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το τι έχει συμβεί σε όλα τα μέρη, σε όλες τις χώρες που ακριβώς ήταν τα προβλήματα και αν υπήρχαν αντιδράσεις από τον τόπιο πληθυσμό, πώς λύθηκε αυτό που οι τεχνικές ήταν επιτυχίες που απέτυχαν. Και με όλα αυτά και σε συντονισμό με την Μητροπομπέλα θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι συστάσεις. Ε, θα πρέπει να δούμε αν θα έχουμε πιο αυστηρό κανονισμό ή όχι. Είμαστε σε αρχικό στάδιο των διαδικασιών και αυτή τη στιγμή εξελίξεις για το συστηματικό αέριο ε, δεν είναι σαφής ακόμη και στην Πολωνία ε, είδαμε ότι υπάρχει μείωση των εγκαταστάσεων υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που εργάζονται από αυτών των θεμάτων που προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι όλες οι περιβαλλοντικές μελέτες εκδικτύπου θα είναι καλής ποιότητας. Αυτά, Πρόεδρε. Σας κατευχαριστούμε για τις λεπτομερείς σας απαντήσεις. Αρχίζει ο δεύτερος γύρος. Πρέπει οι ομιλητές να περιοριστούν στο 1,5 λεπτό. Έχουν ήδη ζητήσει το λόγο 25. Η κυρία Γκαρντίνη πρώτη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε Θέλω να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση για το σύστημα εμπορία εκπομπών που έχει να κάνει με μια συνεχή ανησυχία μου γιατί η οδηγία για τις ΙΕΣ δίνει στα κράτη τη δυνατότητα να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν ε, ε, τα όσα προκύπτουν από τις δημοπρασίες ε, προαιρετικά. Αυτό όμως δημιουργεί στρεβλώσεις. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω εφόσον προκειμένου να μεταρρυθμιστεί το σύστημα ότι Εσείς δεν πιστεύετε ότι ο στόχος της οδηγίας σε ό,τι αφορά τη χρήση των όσων αποκτούνται από τους διαγωνισμούς να χρησιμοποιούνται έτσι ώστε για να υποστηρίξουμε το έμεσο κόστος κυρίως στις βιομηχανίες και στους κλάδους που θίγονται περισσότερο από τη διαρροή του άνθρακα. Ευχαριστώ, Ματίας Γκρότε. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, είσαστε στην Πολωνία την προηγούμενη εβδομάδα και για την Ενεργειακή Ένωση τοποθετηθήκατε και για τον συνολικό κλιματικό στόχο στοιχείο πυρήνα για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία του Περιβάλλοντος και πολιτική με την, το σύστημα εμπορίας τρίπον. Τα συμμερίζομαι όλα αυτά. Ένας πολύ μικρό τομέα στον τομέα των ε, εκπομπών ρήπων και εμπορίας εκπομπών ρήπων έχουμε που μας δημιουργεί πρόβλημα είναι οι διεθνείς αεροπορικές ε, ε, συνδέσεις και μεταφορές και γίνονται διαπραγματεύσεις σε σχέση με την ε, ΑΙΚΑΟ και η ερώτησή μου είναι πώς έχουν προχωρήσει αυτές οι διαπραγματεύσεις ποια είναι η δική σας εκτίμηση για την πρόοδο αυτών των διαπραγματεύσεων εκεί λένε κάποιοι ότι πρέπει να σταματήσουμε το χρονόμετρο εμείς οι Ευρωπαίοι και Άλλοι λένε όχι, είναι η τελευταία φορά κατά την οποία υπήρξε μια ας το πούμε καθυστέρηση. Γι' αυτό με ενδιαφέρει να μου πείτε ποια είναι η δική σας εκτίμηση για την κατάσταση των πραγμάτων και την πρόοδο των διαβουλεύσεων. Και για το offset δεν μπορεί να είναι λύση για τη συμπερίληψη των εναέριων μεταφορών στη στρατηγική μας για την προστασία του κλίματος. Εμείς χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικότερο, αποτελεσματικό μέσο και αποφασίσαμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι το σύστημα εμπορίας τρύπων. Όμως, σε διεθνείς διαπραγματεύσεις καταδείχθη ότι είμαστε ανοιχτοί για την επίτευξη διεθνών λύσεων, αλλά πρέπει να είναι βιώσιμες και αξιόπιστες. Θέλω να ακούσω την εκτίμησή σας για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, καλό σας βράδυ. Η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει και έδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση το σθένος να επιτύχει μια διεθνή συμφωνία πραγματικά δεσμευτική σε σχέση με την ε, συμφωνία για τις ε, κλιματικές αλλαγές στο Παρίσι κατά τέτοιου έτους. Ο τομέας των μεταφορών 25% σε σχέση με τι τις εκπομπές ρήπων θερμοκηπίου Παρ' όλα αυτά όμως σε σχέση για την αντιμετώπιση κάποιων ε, εκπομπών ρήπων από ορισμένους τομείς, ε, ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών δεν έχει ρυθμιστεί τελεσίδικα, εκπέμπονται υψηλές ε, τιμές ρήπων και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μια συνολική τώρα αντιμετώπιση των εκπομπών ρήπων στις θαλάσσιες διεθνείς μεταφορές έχει πολύ μεγάλο ρόλο και έχει και μια προοπτική ας το πω έτσι διάρκειας 10 ετών στην ε, Ολομέλεια θα εγκριθεί ένα σύστημα για την ε, ταυτοποίηση και κωδικοποίηση των εκπομπών ρήπων για τις θαλάσσιες μεταφορές η ερώτηση είναι η εξής επίτροπε θεωρείτε ότι θα υπάρξει μια διεθνής αποδοχή αυτού του συστήματος ή όχι. Δεύτερη ερώτηση. Ποιε είναι οι δικές σας προσδοκίες για να υπάρξει πρόοδος. Πρόοδος στο επίπεδο του, διεθνού Διεθνούς Θαλάσσιου Οργανισμού σε σχέση με το πρωτόκολλο των Παρισίων. Τρίτη ερώτηση. Θεωρείτε ότι ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών θα αποφύγει να εγγραφεί, να ενταχθεί στο ε, σύστημα των ε, εκπομπών ρήπων και τι θα πρέπει να γίνει μέχρι τη συμφωνία αυτή ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία στο Παρίσι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα η κυρία Τόρες Ματίνες παρακαλώ. Ευχαριστώ ιδέα ότι μπορούμε να σώσουμε τον κόσμο τελευταία στιγμή και να πολεμήσουμε τον χρόνο σημαίνει της ταινία. Αυτό ισχύει και για την κλιματική αλλαγή. Ε, αυτό που κάνουμε σήμερα θα καθορίσει το αύριο. Ο καρπός της συμφωνίας του Δεκεμβρίου στο Παρίσι θα πρέπει να πετύχει το στόχο της ε, μείωσης ε, ε, των δύο βαθμών. Κυρία Κανιέτε, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα περικόψει τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου χωρίς να μειώσει την χρήση των ορυκτών καυσίμων, γιατί από ό,τι βλέπουμε και μέσω της υδραυλικής ρογμάτωσης αυξάνουμε την εξόριξη αυτών των καυσίμων και επίσης η Ευρωπαϊκή ε, η Ισπανική κυβέρνηση τι λέει για αυτό που έγινε στα Κανάρια την περασμένη εβδομάδα. Τώρα εδώ αποφασίζουμε για το μέλλον της γης και της ανθρωπότητας, οπότε είναι πολύ σημαντικό. Thank you very much. And now... Ευχαριστώ κύριε Γιάπα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχω τρία ερωτήματα και αν ξεπεράσω χρόνο θα με σταματήσει ο πρόεδρος. Πρώτον, η ενεργειακή αποδοτικότητα. Κύριε Κανέτε μου, είπατε ότι ένας από τους στόχους είναι να εφαρμοστεί η οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα και συμφωνώ ότι η εφαρμογή της θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό γιατί τρία χρόνια μετά από τη θέση ενισχύ της οδηγίας αυτής 27 από τα 28 κράτη-μέλη ερευνώνται από την Κομισιόν, διώκονται από την Κομισιόν γιατί δεν την εφάρμοσαν και η χώρα μου είναι μέσα σε αυτές. Υπάρχει νομοσχέδιο στον Κρικό Κοινοβούλιο για να διορθωθούν τα πράγματα αλλά δεν είναι ψευδολύση. Νομίζω λοιπόν ότι η Κομισιόν κάνει λάθος στην εκτίμηση της της δράσης των χωρών μελών και της προόδου των διότι η οδηγία δεν έχει εφαρμοστεί γιατί σαμποτάρεται από τα κράτη-μέλη. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι ως το 20 ή και μετά το 20 αφού δεν έχουμε ακόμη καν δεσμευτικούς στόχους για το μετά το 20. Μόνο ευσεβείς Πόθη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πέτρελε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τα σαφή σας λόγια και την φιλόδοξη σας προσέγγιση. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο συμφώνησαν να αυξηθεί στο 27% η ενέργεια χωρίς διοξίδιο. Συμφωνώ ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πρέπει αυτές να είναι το 27% θα είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους αλλά για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πρέπει νομίζω να έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Ερωτώ λοιπόν, τι έχει αναλυφθεί από την Κομισιόν για να δημιουργηθεί μια τέτοια γενική στρατηγική για όλους τους τομείς, ιδιαίτερα ενδιαφέρομαι για την συνεργασία μεταξύ θεμάτων περιβάλλοντος, ενέργειας και κάτι άλλο. Ελπίζω μαζί με τα κράτη-μέλη να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο επενδύουμε τα δημόσιο χρήμα για τη στρατηγική μεταξύ άλλων των ενεργειακών στόχων 2030. Υπάρχει η έννοια των εξύπνων πόλεων αλλά χρειάζονται και η έξυπνη ύπεθρος χρειάζεται. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξουν έξυπνα πλαίσια με μία ενιαία στρατηγική. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ μου. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρέπει να στεφτεί με επιτυχία το εγχείρημα. Ερώτημα για σας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι σημαίνει επιτυχία στο Παρίσι, ποιο πρέπει να είναι το αποτέλεσμα για να θεωρηθεί επιτυχία. Έχουμε τη διπλωματία για τα κλιματικά θέματα που ξεκίνησε με την Πολωνία και άλλες ε, χώρες. Θα έχουμε και μια συνάντηση με την Κίνα που έχει προγραμματιστεί, μια ξεχωριστή πρωτοβουλία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας ε, για το Παρίσι όπως ε, το έκαναν και οι με την Κίνα πέρυσι. Υπάρχει ένας μεγάλος ε, τομέας ε, εκπομπών ρήπων που είναι οι αλλογενοποιημένες εκπομπές ρήπων Υπάρχει πρόοδο σε σχέση με αυτό το θέμα όπως είδαμε στην διάσκεψη της ε, Μπανκόκ. Είναι σημαντικό στο πρωτόκολλο του Μοντρεάλ να ενταχθούν αυτά, αλλά θα πρέπει να αναλάβει μια ομάδα κρατών την πρωτοβουλία για κάτι τέτοιο. Έχει λοιπόν ε, ε, υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μοντρεάλ για την ε, ευρωπαϊκή, τον ευρωπαϊκό ε, προεκλογικό αγώνα όσον αφορά τις ηλεκτρικές συσκευές ε, μπορούμε να είμαστε πολύ αποτελεσματικότεροι και να είμαστε πολύ πιο αποδοτικοί στην εκμετάλλευση της ενέργειας επειδή υπάρχει τεχνολογική πρόοδος για αυτές τις συσκευές. Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάμπους. Καταρχήν, θα σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας Επίτροπε και για την σπουδαιότητα για την συμμετοχή σας η διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρεις ερωτήσεις πολύ σύντομες. Η πρώτη για τη διακυβέρνηση στα τέσσερα επίπεδα, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης. Θα μπορούσατε να εξειδικεύσετε πώς θα πρέπει τα διάφορα επίπεδα μέσα σε ένα κράτος ε, της ε, διακυβέρνησης να ενταθούν στην ενεργειακή διακυβέρνηση. Δεύτερη ερώτηση για την κοινή αγορά αερίου και αναφερθήκατε στο φυσικό υγροποιημένο αέριο Γνωρίζετε ότι σε άλλες περιοχές της Ευρώπης αλλά και, τεχνο... και τη... στην Ισπανία και Καταλωνία έχουμε... υπάρχει αυτή η τεχνολογία αλλά θα πρέπει να υπάρχει διασύνδεση και στις 28 Νοεμβρίου δόθηκε η απάντηση ότι έχει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσει εκ του σύνεγγης ε, την εκτέλεση, την υλοποίηση αυτού του προγράμματος προτού υλοποιηθεί το 2020. Τι γίνεται σε σχέση με αυτή την πρόθεση. Θα είμαστε έγκαιρα, θα έχουμε προχωρήσει μέχρι το 2020 σχετικά μια τρίτη ερώτηση για τα ανανεώσιμα Πολύ σύντομη ερώτηση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή Επίτροπε. Υπάρχουν πολιτικές στα κράτη-μέλη που φαίνεται ότι δεν πορεύτηκαν προς την κατεύθυνση, την επαρκή κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Συμμερίζομαι τους λόγους για την Ισπανία, για τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν στη χώρα μας, αλλά πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσλειτουργίες. Ή σε επαφή με τα κράτη-μέλη υπάρχει η διαπίστωση από πλευρά σας ότι υπάρχει βούληση να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να απηχήσω τις ευχαριστίες ε, των μελών της Επιτροπής για την παρουσία σας και τα, την τοποθέτησή σας. Μια ερώτηση για τον ρόλο για την Ενεργειακή Ένωση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ενεργειακή αποδοτικότητα πρέπει να εξετάζεται ως κύρια προτεραιότητα για την σταθερή αξιόπιστη ενεργειακή τροφοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά πολλές φορές ε, δεν εντάσσονται τα θέματα της εξόριξης ε, κάποιων ε, ενεργειακών πόρων και υπάρχει η κατάληξη στους εξορίξιμους πόρους και αυτό ε, οδηγεί σε κάποιες ε, επιλογές. Η δική σας θέση για την, ε, τον τομέα αυτό ποια είναι, τι κάνετε σε σχέση με τους συναδέλφους σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί χρειαζόμαστε και την επάρκεια πόρων και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Τι γίνεται λοιπόν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αντιμετωπιστούν τα θέματα για παράδειγμα αποβλήτων και να υπάρξει η ενεργοποίηση όπως απαιτείται στην ορθή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, λέω κύριο Σφαρία, για μια ακόμη φορά επανέρχομαι στις ερωτήσεις. Ε, άμεσα τώρα ο κύριος Τόρβαλτς μου ζήτησε να πάρω το λόγο για αυτόν και θα μιλήσω αγγλικά γιατί έχω την ερώτηση στα αγγλικά. Στην ε, Ενεργειακή Ένωση. Μπορώ και πορτογαλικά, μπορώ, αλλά αγγλικά. Στην ανακοίνωση της 25ης Φεβρουαρίου η Κομισιόν είπε ότι πρέπει η Ένωση να επενδύσει περισσότερο σε εναλλακτικά βιώσιμα καύσιμα. Και γι' αυτό χρειάζονται μακροπρόθεσμα προγράμματα για σταθεροποίηση του επενδυτικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα όμως και για διάφορους άλλους λόγους πρέπει να γίνει αυτή η διαφοροποίηση. Πρέπει να αναρωτηθούμε μήπως οι επενδύσεις καθυστερούσαν διότι δεν ήταν σαφή τα προγράμματα. Ως προς αυτό πώς με την Ενεργειακή Ένωση μπορούμε να πάρουμε μαθήματα από τα παρελθόντα λάθη μας και να έχουμε εκ των προτέρων λύσεις. Ευχαριστώ. Thank Κυρία Τάλη, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε που μας επισκέπτεστε τόσο τακτικά για να μας ενημερώνετε. Φαίνεται ότι υπάρχει ευρεία συνένωση ότι ένα σωστά ρυθμισμένο ETS μπορεί να μας βοηθήσει για την αντιμετώπιση και των κλιματολογικών αλλαγών και νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει και με τη συμπερίληψη περισσότερων παραγόντων. Πώς νομίζετε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον το ETS το πρόβλημα πολλών τομέων ως προς τις εκπο... των εκπομπών διοξιδίου. Αν θέλετε να επεκτείνετε το ETS, ποιους τομείς θα συμπεριλάβει το μέλλον. Thank you very much. Now, Mr. Ο κύριος Εκ. Yeah, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για αυτή τη συζήτηση που έχουμε και σας ευχαριστώ και για την πολιτική που ακολουθήσατε για το κλίμα και χαιρετίζουμε όλες σας τις προσπάθειες ώστε η διάσκεψη κορυφής στο Παρίσι για το κλίμα να στεφθεί με επιτυχία. Αλλά για να είμαι ειλικρινής είχα υπόψη να είχαμε πιο φιλόδοξους στόχους η μείωση των υπομορήπων μέχρι το 2050 θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη πιστεύω εδώ. Αλλά η ερώτησή μου είναι γνωστό από επιστημονικής πλευράς ότι παράλληλα με άλλα αίτια και ε, τα ισοδύναμα εκπομπών ε, ε, διοξιδίου του άνθρακα παγκόσμια έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις και θα έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις για το κλίμα μας και γι' αυτό θα πρέπει με ειλικρίνεια ανοιχτά να συζητήσουμε αυτά τα θέματα έχουμε 1,5 δις των ε, ε, στον πλανήτη μας ε, και εκπέμπονται τέτοιου είδους αέρια και επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα και σύμφωνα με διεθνείς μελέτες η συνολική βιομηχανία κρέατος είναι 18% των, του συνόλου των εκπομπών λοιπόν πέρα από τις ατομικές ή συλλογικές συνδρομές των οχημάτων ή των πλοίων που είναι 40% συνολικά. Ερώτησή μου, αυτό το ζήτημα, αυτό το θέμα θα το αναφέρετε στο Παρίσι για τέτοιου είδους εκπομπές ρήπων που μέχρι σήμερα ήταν ταμπού. Θα τα θέσετε επί σε αυτά τα θέματα. Θα με ενδιέφερε η άποψή σας γι' αυτό. Θα τοποθετηθείτε στο Παρίσι επ' αυτού του προβλήματος. Θα προσπαθήσετε κάτι να αλλάξετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μποναφέ. Καλησπέρα σας και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και για τις απαντήσεις σας είναι πολύ ακριβή. Εγώ τώρα θέλω να πάω στο Παρίσι πολύ σύντομα, γιατί πιστεύω ότι και τι επόμενε εβδομάδε ε, τα μάτια του κόσμου λέει και ελπίδε ε, θα είναι στραμμένε ε, στην COP21 και εσεί και οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων έχουν μεγάλη ευθύνη να ελοποιήσουν μια συμφωνία φιλόδοξη, καθολική και δεσμευτική και δεν θα αρκέσει γιατί φυσικά δεν αρκούν οι συμφωνίες, ε, πρέπει κατόπι να τις θέσουμε και σε εφαρμογή. Από τη σκοπιά αυτή ήδη εμ, υπογραμμίστηκε ότι είναι πολύ σημαντικές οι επενδύσεις, όχι μόνο οι δημόσιες, ε, ίσως να μην αρκούν, αλλά και οι ιδιωτικές και οι ιδιώτες παρακολουθούν πολύ προσεκτικά το πώς εξελίσσεται τη συζήτηση γύρω από τη διάσκεψη των μερών 21 και ο χρόνος εφαρμογή συμφωνίας και φυσικά η νομική φύση της συμφωνίας και το πιο γεωγραφικό εύρος θα πάρει. Θα βαρύνουν όλα αυτά στις επιλογές των επενδυτών. Όμως, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ε, Πόσο στην Ευρώπη σκεφτόμαστε να εκμεταλλευτούμε τις ιδιωτικές επενδύσεις και σε σχέση με το σύνδιο Juncker μπορούμε να σκεφτούμε να δημιουργήσουμε ένα μέσο ad hoc πλατφόρμες ειδικέ παραδείγματος χάρη για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και πώς σκέφτεστε να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως ε, το ε, Green Carbon Fund των Ηνωμένων Εθνών, αυτό το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ κύριο Σλέκ. Ευχαριστώ. Και εγώ χαιρετίζω τον Επίτροπο. Ακούσαμε μερικά αντιφατικά πράγματα από την Κομισιόν. Από τη μία ο Επίτροπος μιλά για φιλόδοξα στόχους αντιμετώπισης των κλιματολογικών αλλαγών. Απ' την άλλη όμως ακούμε ότι εξαρτώμαστε ακόμα πολύ από τον άνθρακα διότι έχει το δικαίωμα κάθε κράτος να καθορίσει το ενεργειακό του λέει μείγμα. Πριν από τρεις μέρες ο αντιπρόεδρος Σέλσεβιτς στο Βελιγράδι μίλησε για τις ανανεώσιμες και για βιώσιμες πηγές ενεργείας και είπε ότι έτσι θα μπορέσουμε να γίνουμε παγκόσμιοι ηγέτες και να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το πετυρέλαιο. Η Ιταλία και η Κροατία δε, απ' την άλλη, ψάχνουν για κοιτάσματα στην Αδριατική, καθώς και το Μαυροβούνιο και η Αλιβανία. Ενεργειακό μείγμα δεν είναι το θέμα εδώ, αλλά το γεγονός ότι οι χώρες αυτές μιλούν ακόμη για κοιτάσματα ορυκτών υδρογονανθράκων. Αυτά έχονται σε μεγάλη αντίφαση με αυτά που μας είπε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Επικεφαλής της Ενεργειακής Ένωσης. Και με τον υπεύθυνο για την Ενεργειακή Ένωση όπως ξαναείπα και πριν. Λοιπόν, Πώς θα πείσει λοιπόν τις υποψήφιες χώρες και τις χώρες μέλη να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης όπως ανέφερε ο Επίτροπος Έλσονβιτς να μειώσουν δηλαδή το μερίδιο των ορυκτών υδροκοτρανθράκων στο μείγμα τους και πώς θα τις πείσει, πώς θα τις πείσει να χρησιμοποιούν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ κυρία Κάλενμπαχ. Ευχαριστώ θερμά. Πληθώρα ερωτήσεων έχουν κατατεθεί προς εμάς. Δύο θέλω να συμπληρώσω σε δύο σημεία όπως ο Γιώ Λάινερ πιο πριν. Όπως το είπε και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα ότι τον τομέα της οδηγίας ε, για το eco-design, το οικολογικό σχεδιασμό θέλετε να τον προωθήσετε ώστε να υπάρχει καλύτερη προσέγγιση των πολιτών και στην προεκλογική εκστρατεία αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που λαϊκίστικα και αρνητικά με την υπερρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιβαρύνθηκε. Με ενδιαφέρει η επικοινωνιακή σας στρατηγική γι' αυτό. Το θεωρώ ένα από τα σημαντικότερα θέματα, ουσιοδέστερα θέματα για τα θέματα ενέργειας. Δηλαδή πώς θα μπορέσουμε με τον φθηνότερο τρόπο να προχωρήσουμε. Δεύτερη ερώτηση, άσχετα αν αυτό δεν είναι άμεσος τομέας αρμοδιοτήτων σας, υπήρξε ευρύτερο θέμα για τους hacker είναι όχι μόνο ένα πραγματικά ε, πάρα πολύ σημαντικό θέμα που ε, καταλήξαμε στην αυστηρή ερώτηση κατά πόσον εσείς ως Επίτροπος για τα ενεργειακά θέματα σε σχέση με την Ενεργειακή Ένωση μπορείτε να εμπλακείτε σε θέματα ε, διασφάλισης της τροφοδότησης με εναλλακτικά δίκτυα όταν υπάρχουν και δυνατότητες αυτή η ευαίσθητη ε, πλευρά των υποδομών από επιθέσεις hacker τουλάχιστον ε, για κάποιο χρονικό διάστημα να πάψουν να λειτουργούν ή να αδρανοποιηθούν. Πώς θα το αντιμετωπίσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Καμπεσόν. Πρόεδρε. κυρία κανιέτα τα είπατε σχεδόν όλα, αλλά θα ήθελα να επιμείνω σε κάποιες ιδέες που ακούστηκαν απαλλαγή από τι ανθρακούχε εκπομπέ και καταπολέμηση τη ε, κλιματική αλλαγή. Ε, από ό,τι φάνηκε, πολλοί συμφωνούν ε, και αυτό θα γίνει και μέσω της χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών ε, ενέργειας. Όμως ε, ε, βλέπουμε ότι και η αποθήκευση του άνθρακα είναι μια πραγματικότητα αλλά και η πρόσβαση στις ανανεώσιμες πηγές είναι κάτι που θα επιτευχθεί από την πλευρά των καταναλωτών. Και τώρα έχω την πρώτη ερώτηση. Πώς βλέπετε την αναγκαιότητα να προωθήσουμε και να ρυθμίσουμε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν ε, την αυτοκατανάλωση και το θέμα των συνεταιρισμών που επίσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το είδος πολιτικής για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής και δεύτερον είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε αλλαγή στη λειτουργία της ηλεκτρικής αγοράς, της αγοράς ηλεκτρισμού και πρέπει να διευκολύνουμε και τις επενδύσεις σε ανασυρώσιμες πηγές ενέργειας. Ίσως ένας πιο φιλόδοξος ε, στόχος ε, θα ήταν να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στην αγορά και στους επενδυτές και ελπίζω ότι τα αποτελέσματα ε, της διάσκεψης του Περισσίου να μην μείνουν κενό γράμμα από την πλευρά των κρατών μελών με όριο το 2030. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέλετ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα. Κύριε Επίτροπε, δεν θα θέσω ερώτηση για τον ελέφαντα εδώ στην αίθουσα, δεν αναφέρθηκε ακόμη αυτό που είναι το MSR, το αποθεματικό ε, σταθερότητα τη αγορά. Έχουμε και ένα σημαντικό τριμερή διάλογο την επόμενη εβδομάδα και ελπίζω ότι τα κράτη-μέλη ε, σκοπεύουν στο να υπάρχει μια σαφής εντολή και αυτό είναι πολύ κοντά στη θέση και του Κοινοβουλίου. Και δεν αφιβάλλω, κύριε Πίτροπε, ότι και εσεί εργάζεστε προ την διακατεύθυνση με το Κοινοβούλιο. Τώρα έχω συγκεκριμένη ερώτηση για το σύστημα εμπορία εκπομπών. Γιατί φυσικά είναι ένα από του ε, παράγοντε επιτυχία ε, τη διάσκεψη του Παρισιού είναι το ETS. Και ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει μία ε, μεταρρύθμιση του συστήματος έτσι ώστε να καταστεί πιο σταθερό. Και η πιο ιδανική κατάσταση είναι να σχετίσουμε το σύστημα της Ευρώπης με τα υπόλοιπα ETS παγκοσμίω και ίσως να το συνδέσουμε με αυτό της Ελβετίας, αυτό που είναι το πιο κοντινό μας. Έχετε συγκεκριμένα σχέδια λοιπόν της Κομισιόν ε, σε σχέση με τη σύνδεση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών με το Ελβετικό. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, κύριε Πίτροπε, σας έθεσαν πάρα πολλές ερωτήσεις. Έχετε και το χρόνο να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Καρδίνη. Κυρία Καρδίνη. Η κυρία Γκαρδίνη εξέφρασε κάποιο μέλημα, μια, μια ανησυχία, ποια είναι η θέση, είπε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη αυτή τη δυνατότητα εναρμονισμένες ε, πολιτικές να είναι θερκτικές όταν ε, υπάρχουν σημαντικές τεχνικές και τεχνολογικές ε, προκλήσεις διότι τέτοιες συμφωνίες εξαρτώνται από τα όσα είναι διαθέσιμα για τις επιχειρήσεις και ένα μεγάλο ποσοστό για τον επιμερισμό θα αφαιρεί το. Και έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα όσον αφορά το περιεχόμενο εκπομπών άνθρακα που κυμαίνεται πολύ σημαντικά, υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ περιφερειών και αυτό το καθιστά δύσκολο να υπάρξει ένας εναρμονισμός των αγορών. Γι' αυτόν τον λόγο τον Οκτώβριο αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες ότι θα πρέπει να συνεχιστούν αυτά τα μέτρα και με βάση αυτή την προσέγγιση θα μπορέσει να δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πρέπει να γίνει ώστε να αποφευθούν οι στρεβλώσεις στην αγορά ε, λόγω των ενισχύσεων που θα μπορούν να τύχουν κάποιες επιχειρήσεις ενώ κάποιες άλλες όχι σε σχέση με τις δράσεις των κρατών μελών. Θα δούμε λοιπόν την εικόνα αυτή και θα πρέπει να ε, έχουμε υπόψη ε, τις δυσκολίες επίλυσης αυτού του προβλήματος. Όσον αφορά τώρα ε, the ε, ε, τα προβλήματα των διεθνών αεροπορικών μεταφορών πρέπει να σημειωθεί πρόοδος το 2016 σε αυτό το πεδίο. Διαφορετικά θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη κατάσταση αν δεν γίνει αυτό. Στην Ευρώπη συνολικά πρέπει να ληφθούν αποφάσεις λοιπόν και πρέπει να γίνουν συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο για το ποια οδό θα ακολουθήσουμε. Το καλύτερο πιθανό δυνατό σενάριο είναι να σημειωθεί πρόοδος και να μπορέσουν όλοι να ευθυγραμμιστούν σε διεθνές επίπεδο. Το ίδιο γίνεται και για τον Διεθνή ε, Οργανισμό ε, για την Θάλασσα. Και αυτό προσπαθούμε να διεθνή ναυτιλιακό οργανισμό αποστέλλεται ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για τη συνάντηση τον Μάιο στο Λονδίνο και για τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών το Δεκέμβριο στο Παρίσι. Εναίδιες μεταφορές λοιπόν και θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να απηχούνται και να αντανακλώνται στην Συμφωνία των Παρισίων. Για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα πρέπει οι πηγές, τα αίτια της δημιουργίας των προβλημάτων να αντιμετωπιστούν σφαιρικά όλα ολοσχερός ε, από όλες τις πηγές και έτσι λοιπόν θα πρέπει να έχουμε και τις ε, ε, εκπομπές τρύπων από όλες τις πλευρές. Στο πρωτόκολλο κάποια πρόοδος έχει επιτευχθεί. Οι Αμερικανοί και με την παρόμοια, α το πω δράση τους που πρέπει να δούμε τροπολογίες ή τροποποιήσεις από α, χώρες που κατατίθενται που μπορούν να περιπλέξουν την υπόθεση. Στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ θα πρέπει να μπορέσουμε να δούμε αν υπάρχει υποστήριξη για να υπάρξει πρόοδος. Θα είναι σημαντικό να υπάρξει συνεργασία της Σαουδικής Αραβίας <clears throat> και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σε σχέση με τη χώρα αυτή η πρότασή μου λοιπόν είναι να έχουμε πολυσχηδείς επαφές για να μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουμε. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει για τα καύσιμα και τις πηγές ε, τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν το μείγμα, ενεργειακό μείγμα που επιθυμούν. Πρέπει όμως να σέβονται και τους στόχους μείωσης εκπομπών ρήπων που ε, θεσπίζονται τομεακά και σφαιρικά. Υπάρχουν στόχοι λοιπόν που η αποδοτικότητα ενέργειας και ε, οι δράσεις μας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη. Το πραγματικό πρόβλημα θα είναι η διακυβέρνηση. Αν είμαστε σε θέση να ε, θεσπίσουμε ένα πλαίσιο διακυβέρνησης που θα είναι λειτουργικό, και θα είμαστε αποτελεσματικοί, τότε είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη με ομοσπονδιακή δομή, για παράδειγμα, ή με αυτονομία περιοχών και περιφερειών, πρέπει να δημιουργήσουν ένα σύστημα ώστε οι υπεύθυνοι επιτύπου, επιτόπου περιφερειακά και τοπικά να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσει του. Ε, δεν είναι μόνο τα οι κεντρικές αρχές ενός κράτους αλλά και οι τοπικέ και περιφερειακές αρχέ. Όμω ε, οι εθνικέ στρατηγικέ, μια και είναι εθνικού χαρακτήρα, πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα διαλόγου που θα θεσπιστεί για να μπορέσουμε να δούμε πώ θα επιτευχθεί οι στόχοι αυτοί να μπορούν να επιτυγχάνονται μέσα στο περιφερειακό και τοπικό πλαίσιο στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένα περίπλοκο εγχείρημα. Οι μεταφορές ε, ε, που αναφέρθηκε και για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των μεταφορών αποφασίσαμε να τα αντιμετωπίσουμε σε τομεακά ξεχωριστά θα θεσπιστούν για τα οχήματα, τα ΙΧ για παράδειγμα, εκπομπές report, θα έχουμε μια σφαιρική, ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η προσέγγιση για τη μείωση εκπομπών report στις μεταφορές δεν είναι μόνο η μείωση των εκπομπών ε, ανάλογα με την ταχύτητα που ακολουθεί οδηγώντας ο οδηγός ενός γιοταχή. Είναι ένα πολύ πιο περίπλοκο θέμα διαχείρισης ροών, ε, μεταφορών ε, στις πόλεις. Υπάρχει και το θέμα της κοινή προσπάθειας των επιτρόπων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να υπάρξει μια σφαιρική προσέγγιση αντιμετώπισης αυτών και για τα καύσιμα επίσης καθώς επίσης ε, και την, ε, την ασφάλεια που πρέπει να δημιουργηθεί για τους επενδυτές ε, σε ένα πλαίσιο το οποίο θα ισχύει μελλοντικά. Όλα αυτά τα στοιχεία με όλες αυτές τις παραμέτρους στις, στο νομοθετικό πλαίσιο για τα κάψιμα όλα αυτά θα πρέπει να αναθεωρηθούν για την περίοδο 2020-2030 και πρέπει να γίνουν αυτά όλα αρκετά νωρίτερα πριν από το 2020 ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί μια ασφάλεια προγραμματισμού και σχεδιασμού για τις επιχειρήσεις. Ο κύριος Χάρμπορ έκανε λόγο για την, ε, το θέμα αυτό στο οποίο έχει δίκιο. Η οδηγία που δημιούργησε τα μεγαλύτερα προβλήματα για την ε, ένταξη στα νομικά συστήματα των κρατών μελών ήταν η οδηγία για τα ενεργειακά θέματα και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Γι' αυτόν τον λόγο αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει να καθελκύσει όλες τις ε, διαδικασίες ώστε να είναι όλες έτοιμες και να λειτουργήσουν σωστά αναλύουμε ανακράτος τι γίνεται σε σχέση με τη συμμόρφωση και την ευθυγράμμιση με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Να δούμε δηλαδή τι γίνεται σε σχέση με το συγκεκριμένο όριο ή ε, ανόφλη που έχει, κατόφλη που υπάρχει. Από την άλλη πλευρά συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και δίνουμε συμβουλές, συμβουλεύουμε τα κράτη-μέλη πώς μπορούν να υλοποιήσουν ε, τους στόχους αυτούς. Στόχος μας δεν είναι να επιβάλλουμε κυρώσεις στα κράτη-μέλη. Στόχος μας είναι να μπορέσουν να ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, όταν ένα κράτος ε, μέλος έχει ε, κάποια προβλήματα τότε θα πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη σε σχέση με άλλα που δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Επίσης μια παρέμβαση που με, ε, ρωτούσε πώς η στρατηγική για τα ανανεώσιμα θα διαμορφωθεί. Θα υποβάλουμε, θα καταθέσουμε. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εκπονήσουμε ένα έγγραφο, ένα έντυπο πολιτικής με συγκεκριμένες προτάσεις για αυτή την πολιτική τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον ώστε να είναι προπομπός, πρωτοπόρος παγκόσμια ο πρώτος, ο πρωταθλητής. Θα υπάρξει αυτό το έγγραφο στρατηγικής ώστε να συμπεριλαμβάνονται τομεακά σε κάθε επίπεδο όλα τα στοιχεία ώστε να υπάρξουν οι υποδομές, τα συστήματα υποστήριξης και συνδρομής και νοτομίας. Εφόλων αυτών πρέπει να προχωρήσουμε με τον πιο σωστό τρόπο για να γίνουμε παγκόσμιοι πρωτοπόροι, πρωταθλητές. Τώρα, τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει, είναι σαφές ε, ότι ξεκινώντας διαπραγματεύσεις έχει κανείς κάποιο στόχο και κάποιος ανέφερε και είπε ότι το τελευταίο λεπτό δεν είναι δυνατό να σωθεί η, ε, το όλο εγχείρημα. Δυστυχώς ε, στις περισσότερες φορές το τελευταίο λεπτό είναι πολλές προτάσεις που εξετάζονται και αντιμετωπίζονται. Έχουμε πολλές φορές προτάσεις που δεν είναι λειτουργικές. Στο Παρίσι πρέπει να καταλήξουμε σε μια λογική αποτελεσματική συμφωνία. <clears throat> Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν 100 σελίδες ε, που να περιγράφουν ε, όλα αυτά για να μην υπάρχουν 100 προβλήματα στο τέλος. Πρέπει να σημειωθεί πρόοδος πριν από αυτό το επίπεδο στο Παρίσι. Τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έχει ένα πρωτόκολλο, ένα δεσμευτικό όργανο, ένα δεσμευτικό εργαλείο. Δεύτερον, ένα μακροπρόθεσμο στόχο. Γιατί όλα αυτά. Γιατί πρέπει να καθορίσουμε ποια είναι η πορεία μας, να χαράξουμε την πορεία μας. Να πούμε, ορίστε, αυτό θα γίνει από το 2010 μέχρι το 2020 για τις εκπομπές ρήπων και τα Τρίτον, μια δυναμική διαδικασία δραστηριοποίησης με διαφάνεια και λογοδότηση στη διακυβέρνηση για να υποπτεύουμε το τι τεκταίνεται, το τι γίνεται για να μπορούμε να σταθμίζουμε και να αξιολογούμε τις επιπτώσεις και μετά έχουμε επίσης αυτές τις διαστρωματώσεις ένα χρηματοοικονομικό πακέτο μέτρων, μια δέσμη μέτρων για την, ε, τα μέτρα που χρειάζονται να καλυφθούν, που πρέπει να καλυφθούν και θα δούμε τι λειτουργεί και τι προχωρεί και θα έχουμε μια βάση για αυτή τη διαπραγμάτευση. Φυσικά θα κινητοποιηθούν κάποια πράγματα, αλλά διαφάνεια, λογοδότηση και ε, ε, ενεργοποίηση είναι θεμελιώδη σημασία. Σημασίας. Αν ξεκινήσουμε την αναθεώρηση το 2025 για τους πιο φιλόδοξους στόχους και για την, ε, το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών θα δούμε Ποιες χώρες κάνουν τι. Αυτό που επιθυμούμε α, ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι 198 χώρες ε, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να μπορέσουν να ενταχθούν και να συμφωνήσουν και να προχωρήσουν και για να υπάρξει χρηματοδότηση, υποστήριξη για προσαρμογές θα πρέπει να υπάρχει και μεταφορά τεχνογνωσίας για να γίνει αυτό πρέπει να έχει υπάρξει ε, κύρωση μιας ε, ε, συνθήκης, μιας σύμβασης και να δούμε τι θα συνεπάγονται όλα αυτά για όλους. Φυσικά οι ανεπτυγμένες χώρες όντας ένα υψηλότερο επίπεδο θα είναι σε διαφορετική θέση. Δεν θέλουμε όμως να υπάρχει διαφοροποίηση, δια, διαφορετική αντιμετώπιση αναπτυσσόμενων χωρών. Για τη Βραζιλία για παράδειγμα, η, ε, δεν είναι το ίδιο η Βραζιλία όπως το Μαλάουι και δεν μπορεί ισοπεδωτικά να αντιμετωπιστούν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Η μόνη αναπτυσσόμενη χώρα, για παράδειγμα η Γκαμπών στην Αφρική και το Μεξικό που στο παράτημα 2 έχει ενταχθεί, υπάρχει όμως σημαντική διαφορά από το 1990 σε σχέση με την ε, αντιμετώπιση των αναπτυσσόμενων χωρών. Η Κίνα για παράδειγμα που είναι σε θέση πολλά να πράξει ή η Βραζιλία είναι μίζονες οικονομίες παγκόσμια αυτές οι χώρες και για την ε, αντιμετώπιση των κλιματολογικών προκλήσεων, κλιματικών προκλήσεων παγκόσμια πρέπει να τύχουν ξεχωριστής αντιμετώπισης. Λοιπόν, τι θα μπορούσε να γίνει. Οι διαπραγματεύσεις θα είναι δυσχερείς. Πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Όλοι θα πρέπει να ε, ε, αναλάβουν δεσμεύσεις. Υπάρχουν κάποιες χώρες που δεν θέλουν μακροπρόθεσμες, μακρόχρονες δεσμεύσεις ε, και λένε ότι πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση. Είναι δύσκολα λοιπόν τα πράγματα, περίπλοκα. Στο τέλος θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα συμπεράσματα και πώς θα προχωρήσουμε και ένα ε, σχέδιο οικολογικής προσέγγισης ή ε, οικολογικού σχεδιασμού. Τι θα γίνει με τα σύμβολα, τα λογότυπα. Ένα οικολογικό τέτοιο σύμβολο και για τις νέες συσκευές που διοχετεύονται στην αγορά και είναι πολύ αποτελεσματικές και την, ε, το, το κόστος και την εξοικονόμηση που επιτυγχάνουν είναι πολύ αποτελεσματικές και εξοικονομούν και χρήματα για παράδειγμα. Το θέμα αυτό πρέπει να το δούμε λοιπόν ενεργά. Και το θέμα είναι το θέμα των αγορών, ότι υπάρχουν πολλές συσκευές που είναι υπερήλικες. Αυτό που προτείνουμε σε, και προτείνεται σε κράτη-μέλη είναι να καταλήξουμε να υπάρξει εκπόνηση ενός προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσουν όλες οι συσκευές ε, να μπορέσουν ε, να ε, προσαρμοστούν και να ε, μπορέσουν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια ενεργειακής αποδοτικότητας. Το ίδιο το οποίο κάνουμε και έχουμε κράτη που θέλουν να αντικαταστήσουν όλα τα παλαιά υπερήλικα οχήματα και, δίνουν, οχήματα και δίνουν και κρατικές ενισχύσεις ε, ως πριμ για να μπορέσουν οι πολίτες να αγοράσουν σύγχρονα τεχνολογικά οχήματα για την επιδότηση της αγοράς τους. Μια τέτοια προσέγγιση πρέπει να ακολουθηθεί λοιπόν αν γίνεται για τον κύριο Κάμπος που ανέφερε το θέμα των ε, ε, των προβλημάτων που υπάρχουν ανακράτως ε, για τις κρατικές πρωτοβουλίες και ρυθμίσεις. Αυτό δημιουργεί ένα περίπλοκο θέμα. Αν κάνει το βήμα ένα κράτος μέλος να επιμερίσει τους στόχους ε, για τα ανανεώσιμα ε, στα μεταξύ των περιοχών ή ε, επαρχιών του. Μέχρι σήμερα δεν το έχουν κάνει όλοι και αυτό είναι ένα πιο περίπλοκο θέμα στη συζήτηση. Μπορώ να σας διασφαλίσω ο επιμερισμός των διαφορετικών δράσεων και τα ποσοστά, οι ποσοστώσεις που θα ισχύουν για ένα κράτος μέλος, αν αυτό είναι περίπλοκο, φανταστείτε πόσο περίπλοκο είναι το εγχείρημα αυτό σε μια ευρύτερη κλίμακα. Για τα θέματα του αερίου και του υγροποιημένου αερίου οι δυνατότητες είναι τεράστιες και φυσικά η αεραγωγή με την ε, Αλγερία και η δυναμικότητα που έχουν να τροφοδοτούν την ε, Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία με υγροποιημένο αέριο και έτσι σε σχέση με τον Νότο θα μπορούσε η Γαλλία να συνδέει, να συνδέεται με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Τι γίνεται για παράδειγμα σε σχέση με τις βαλτικές χώρες ε, και με την νοτιοανατολική Ευρώπη, με, τους, ε, τη διασύνδεση αυτών των αγωγών ε, για παράδειγμα που θα, μπορούσε να, να μπορούσαμε να στοχεύσουμε τα εγχειρήματα και τα σχέδια η ηλεκτρικής ε, διασύνδεσης με την Ακητανία και οι δύο διαπυρηναϊκές διασυνδέσεις ε, η ηλεκτρικής μεταφοράς ενέργειας ε, που θα πρέπει μέχρι τα τέλη του έτους να μπορέσουν να ολοκληρωθούν θα πρέπει οι αρχές να μπορέσουν να ολοκληρώσουν αυτό το εγχείρημα μεταξύ των Ισπανικών αρχών των Γαλλικών αρχών και των Πορτογαλικών αρχών ώστε να προχωρήσουμε σε σχέση με αυτό αυτό το θέμα. Για τα ανανεώσιμα είναι αληθεύει ότι υπάρχουν ε, πολιτικές που είχαν επιπτώσεις ε, στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων. Η Ισπανία έχει σημειώσει πολύ πρόοδο σε σχέση με αυτό το επίπεδο και θα δούμε σε σχέση με το 2020 ε, αν είναι δυνατό να επιτευχθεί το 20%, το 20%, το 16,5% ή το 17% θα ήταν εφικτό. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες διασύνδεσης των υποδομών για να υπάρξει ένας εναρμονισμός. Θα επιθυμούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν γίνεται, τα συστήματα αυτών να μπορέσουν να περάσουν από την αγορά και σε πολλά κράτη-μέλη δίνονται μηνύματα εντάσσοντας ένα σύστημα υποστήριξης ε, σε σχέση με τις ε, κρατικές επιδοτήσεις ή ε, πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα. Άλλος Ευρωβουλευτής μίλησε για το θέμα των βιοκαυσίμων και αν είναι δυνατόν να γίνεται αγορά αυτών των βιοκαυσίμων τι θα γίνει με αυτά τα βιοκαύσιμα θα αναθεωρήσουμε το πλαίσιο αυτό για να μπορέσουμε να επιλέξουμε υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε υπάρχει καθορισμός κάποιων ορίων ή ποσοστώσεων μετατροποποιούνται κάποια πράγματα πρέπει να υπάρξει ένα, μια δέσμη μέτρων και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αυτά τα κάψιμα. Θα υπάρχει ένα ε, περιθώριο, έχουμε μια εκτίμηση για το 5% σε σχέση με το 2012 και ένα περιθώριο που υπάρχει για ένα, μια αύξηση αυτού του ποσοστού ε, μέσα σε μια χρονική προοπτική. Ο κύριος ε, Φαρέας τώρα. Είναι σαφές ε, ότι ε, θα πρέπει να προωθήσουμε τις προσπάθειες για τη χρηματοδότηση των βιοκαυσίμων γιατί έχουμε μείνει πίσω τα βιοκαύσιμα της δεύτερης γενιάς έχουν πολύ μικρή πρόοδο, σημειώνουν πολύ αργή πρόοδο και θα πρέπει στο μέλλον να τα χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας για την κλιματική αλλαγή. Κύριο Σέκ. Αναφέρθηκε στο πρόβλημα του τι συμβαίνει με τη γεωργία, με την εντατική γεωργία Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πήρε την απόφαση να κάνει πολλές αλλαγές στην δασοκομεία ε, σε ό,τι αφορά και τον επιμερισμό των προσπαθειών. Και τώρα συζητάμε με τα κρότη μελη πώς θα το κάνουμε με ένα αυτόνομο πυλώνα, πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Αλλά θα έχουμε και κανόνες λογοδοσίας, ε, θα δούμε και πώς αντιμετωπίζει ο τομέας ε, της ε, προκλήσεις ε, του τομέα της δασοκομείας και θα πρέπει να έχουμε πολύ σαφείς μεθόδους υπολογισμού για να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος του γεωργικού τομέα συνολικά. Δηλαδή δεν πρέπει να δούμε μόνο τι συμβαίνει με τα βοηδή και την εντατική εκτροφή τους αλλά θα πρέπει συνολικά να δούμε τι συμβαίνει με τις εκπομπές από τον τομέα της γεωργίας και πώς τις υπολογίζουμε γιατί δεν μπορούμε να πηγαίνουμε μπρος-πίσω. Θέλουμε να συνεργαστεί και ο τομέας αυτό στην επίτευξη των στόχων. Τώρα, για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Πώς ιδιώτες θα συμμετέχουν στη χρηματοδότηση. Έχουμε θεσπίσει την ενεργοποίηση 100 δισεκατομμυρίων ε, δολαρίων μέχρι το 2020 και από η δημόσια και από ιδιωτική χρηματοδότηση και θα δείτε τους υπολογισμούς ε, σε σχέση με το σημερινό επίπεδο χρηματοδότησης που βρισκόμαστε σήμερα. Είμαστε από το 40 μέχρι το 148 γιατί είναι πολύ δύσκολο να υπολογίσουμε και είναι μάλιστα πολύ δύσκολο να υπολογίσουμε την προσαρμογή Δηλαδή, είναι δύσκολο να υπολογίσουμε τι ενεργοποιούν τα κράτη-μέλη για την κλιματική αλλαγή. Όταν πρέπει να υπολογίσουμε τι κάνει ο δυτικός τομέας για την προσαρμογή, πολλές φορές υπάρχουν μεγάλα project, ένα λιμάνι παραδείγματος χάρη και εκεί εντάσσεται και προστασία των ακτών. Ποια είναι η συνιστόσα τώρα της προσαρμογής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπολογιστεί. Όμως η πιο σημαντική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση ιδιωτική χρηματοδότησης για την κλιματική αλλαγή, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, είναι να μην υπάρχει θεσμικός κίνδυνος ε, για ε, το να έχουμε κακό επενδυτικό κλίμα. Θα πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες και γραμμές ε, για τις επενδύσεις ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι πολύπλοκο το πρόβλημα της ενεργοποίησης της χρηματοδότησης. Ο κύριος ε, Σέλα έκανε μια πολύ δύσκολη ερώτηση για τις αντιφάσεις και τι γίνεται με τη χρήση των ερεκτών καυσίμων. Όταν λέω ότι έχουμε δεσμεύσεις φιλόδοξες αρκεί να δείτε ε, τις INDCs ε, που είναι επιτάπητος στις εθνικές καθορισμένες προτάσεις συνεισφοράς. Ρωτήσατε τι γίνεται με την Ελβετία. Η Ελβετία ήταν η πρώτη, αλλά είναι μια μικρή χώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα βλέπετε τους Αμερικανούς, το Μεξικό, το Λίχτενστάιν, Καμπόν, Μεξικό, Νορβηγία μέχρι τώρα. Με τις ένδυσεις που έχουμε επιτάπητος έχουμε φιλόδοξη δέσμευση της ευρωπαϊκής πλευράς. Είναι σαφής ο στόχος. Είναι εσωτερικός γιατί μιλάμε τουλάχιστον για το 40% εγχωρίως. Δεν έχουμε διεθνείς πιστώσεις, άλλοι έχουν. Έτσι λοιπόν κάνουμε μία προσπάθεια εντός της δικής μας επικράτειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Τώρα από την άλλη να πετύχουμε το στόχο αυτό πρέπει να βρούμε μία εξισορρόπηση. Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές 40% αλλά πρέπει να φτάσουμε στο 30% ενεργειακή αποδοτικότητα και 27% για τις ανανεώσιμες. Έτσι λοιπόν, κρατημέλη, πρέπει να χάρη κρατεί η Ιταλία στο ενεργειακό μείγμα τους ή άλλα κράτη έχουν επιλέξει να πάνε προς την τάδε κατεύθυνση, αυτό μπορούν να το κάνουν αλλά θα πρέπει να σεβαστούν και τους στόχους και να μειώσουν τις εκπομπές και σε άλλους τομείς έχουν μια ολόκληρη γκάμα, έχουν παραδείγματος χάρη τη θέρμανση, τη γεωργία, τις μεταφορές, την ψήξη, έχουν τις επιδόσεις των κτηρίων. Έχουμε μια σειρά στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των εκπομπών στα κράτη-μέλη. Πρέπει να θεσπίσουμε ξεκάθαρη διακυβέρνηση για να διασφαλίσουμε ότι θα παρακολουθούμε την πλήρωση των στόχων κατά τη διάρκεια όλης της περίοδου. Και εκεί είναι που πρέπει να κάνουμε σκληρή δουλειά. Κύριος Κάντενμπεκ, αναφέρθηκε στον οικολογικό σχεδιασμό. Είναι μια καλή οδηγία αυτή, όμως ε, είχαν, είχε υπάρξει κριτική σε προκλογές εκστρατείες, στην όλη ιδέα όμως οι καταναλωτές έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο με περισσότερες ε, συσκευές ε, αποδοτικότητας ανά νοικοκυριό τη χρονιά. Αυτό λειτουργεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτάσει στην πρώτη θέση, σε αποκλεισμένη ηγετική θέση, στην κοινοτομία. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να επιλέξει κανείς πολύ προσεκτικά τα νέα προϊόντα. Πρέπει να είναι αποδοτικά και πρέπει φυσικά να δούμε και τι γίνεται με τις οργανώσεις καταναλωτών. Θα πρέπει να έχουμε πολύ καλό διάλογο με τις οργανώσεις καταναλωτών, να επικοινωνούμε, να κοινοποιούμε καλά τα ωφέλη της πολιτικής και να προλαμβάνουμε τις κριτικές. Να λένε α, τι θέλει η Κομισιό να περιορίσει ε, την ισχύ της ηλεκτρικής κούπας. Ε, αλλά ξεχνάνε, παραδείγματος χάρη, ε, τα ψυγεία, τους υπολογιστές, όλα αυτά έχουν βελτιωθεί και η Κομισιόν πολύ προσεκτικά θα επιλέξει τα νέα προϊόντα. Υπήρξε και μια ερώτηση ah, well, of course. In the, in Λοιπόν, για το σχεδιασμό στην ανακοίνωση για το σχεδιασμό της ενεργειακής αγοράς ε, κάτι που θα πρέπει να προσεγγίσουμε είναι η αυτοκατανάλωση, ε, η συμπαραγωγή, η αυτοπαραγωγή και όλα αυτά τα φαινόμενα. Να δούμε πώς εντάσσονται στο δίκτυο και πώς θα διευκολύνουμε την ανάπτυξή τους, ελέγχοντας και κατά νου ότι αυτές οι διαδικασίες ε, πρέπει να είναι τακτοποιημένες, ρυθμισμένες, γιατί το δίκτυο δέχεται, δέχεται και τις ανανεώσιμες πηγές, όπως και τη συμπεραγωγή, την αυτοκατανάλωση και οποιαδήποτε άλλη μορφή παραγωγής και διανομής ενέργειας. Γι' αυτό θα έχουμε ένα κεφάλαιο που θα το αφιερώσουμε στο να σκεφτούμε πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε τα θέματα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι κίνητρα μπορούμε να δώσουμε στα κράτη-μέλη, ποιο είναι το λογικό κόστος ε, για τη διατήρηση του δικτύου. Όταν έχουμε παραγωγή παντά στο δίκτυο έχουμε κάποιες δαπάνες θα πρέπει να καλυφθούν, αλλά δεν θα πρέπει αυτά να είναι τόσο αποτρεπτικά για να μας εμποδίσουν να το θέσουμε στην πράξη. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε στο θέμα αυτό. Υπήρχε και μια ερώτηση για τα Κανάρια. Εγώ ως Επίτροπος να προσπαθώ να, να τοποθετούμε στα θέματα ευρωπαϊκά, όχι στα θέματα της Ισπανίας, γιατί εκπροσωπώ όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Έτσι, λοιπόν, ε, εδώ δεν επιτίθεμαι, ούτε περασπίζω κάποια εθνική κυβέρνηση. Αν ε, δεν σέβεται μία οδηγία, ε, τότε μπορώ να τοποθετηθώ. Η μακρά μου εμπειρία σε ό,τι αφορά τη διαχείριση περιβαλλοντικών κρίσεων, Εξής, όταν υπάρχουν ε, πετρελαιοκυλίδες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και πρωτόκολλα και καθώς είχε πάρα πολλές πετρελαιοκυλίδες η Ισπανία όπως ε, του Πρεστής ε, οι δράσεις πρωτοκολλούνται και αυτό που γίνεται είναι να εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα. Από όσο διαβάζω στον τύπο έχω την εντύπωση ότι εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα όπως πρέπει κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, ε, υπάρχει μια καλή συνεργασία. Όπως πάντα στις περιπτώσεις αυτές ε, δημιουργείται μεγάλη ανησυχία και είναι και λογικό, κρούμε τον κόκκινο του κινδύνου γιατί πρέπει να προστατεύουμε τα οικοσυστήματα. Όμως εγώ προσωπικά ούτε έχω κάποια κρίση συγκεκριμένη, ούτε είμαι και αρμόδιος. Δεν μπορώ να σας απαντήσω ως επίτροπος, ως πολίτης ε, σας απαντώ και ως ε, πρώην υπουργό, ξέρω ότι υπάρχει μια σειρά πρωτοκόλων που πρέπει να εφαρμοστούν. Όμως ε, βλέπουμε και τι πρέπει να συμβεί σε κάθε περιστατικό και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε πιο πολύπλοκα συστήματα και ξέρετε ότι χρησιμοποιούμε ε, και συστήματα για να ανακτήσουμε ένα σκάφος που έχει βυθιστεί παραδείγματος χάρη στα 2.500 μέτρα ρομπότ ή άλλα. Και η τελευταία ερώτηση ήταν για την Ελβετία και τις αγορές. Η επιθυμία θα ήταν όλες οι αγορές του κόσμου να ήταν ολοκληρωμένες Ο στόχος θα είναι να έχουμε μία πλήρη ολοκλήρωση των παγκοσμίων αγορών. Με την Ελβετία έχουμε φυσικές συνθήκες να συνδεθούμε γιατί υπάρχει σύνδεση των συστημάτων μας, όμως τώρα έχουμε κάποια θεσμικά προβλήματα με την Ελβετία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Συζητούμε με την κυβέρνηση της Ελβετίας για να λύσουμε προβλήματα για τους κώδικες των δικτύων και άλλα. Αν ε, τα λύσουμε στη διαδικασία διευθέτησης, Έχουμε κάποια κρεμή ζητήματα αυτή τη στιγμή, αλλά όταν ε, τα λύσουμε, ε, η πρώτη αγορά με την οποία θα μπορούσαμε να συνδεθούμε θα είναι η Ελβετική, θα μπορούσαμε όμως να προχωρήσουμε και με άλλες αγορές. Συνεργαζόμαστε με άλλες χώρες για να ε, προωθήσουμε τα θέματα αυτά. Έχουμε καλή συνεργασία με την Κίνα και τις ΗΠΑ. Και μια άλλη ερώτηση που ξέχασα. θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη δέσμευση και παγίδευση του άνθρακα, γιατί αν μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτή την τεχνική στα επόμενα λίγα χρόνια, ο Άνθρακα θα μπορούσε να παραμείνει στο ενεργειακό μείγμα, χωρίς να αποτελεί εμπόδιο για να πετύχουμε τους παγκόσμιους στόχους για το κλίμα. Το 2050 τώρα έχουμε κατά νου μείωση 40% των εκπομπών για το 2030. Το 2050 ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 60. Και το 2100 είναι 0. Προκειμένου λοιπόν να προετοιμάσουμε το μέλλον και να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την πορεία, θα πρέπει να αναπτύξουμε τεχνικές δέσμευσης και, και αποθήκευσης του άνθρακα, έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε στον ορίζοντα του 2020 να επενδύουμε όσο δυνατόν περισσότερο στην καιροτομία και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο στάδιο του να διατεθεί στην αγορά για να έχουμε επιτυχία σε αυτό το τομέα. Αφιερώνουμε πολλές προσπάθειες σε αυτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Πριν καταλήξουμε, θα ήθελα να μιλήσουμε για την έγκριση των πρακτικών της 29ης Ιανουαρίου και 18ης Μαρτίου, Αν δεν ακουστούν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, τώρα δηλαδή, θα εγκριθούν. Και μετά η επόμενη συνεδρίαση Βρυξέλλες 6 και 7 Μαΐου. Καληνύχτα. Ευχαριστώ un attimo